Shall we go? Thank you all. Thank you all the colleagues. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Thank you all. Good afternoon. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε την τακτική συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Διεξάγεται συνεδρίαση μέχρι αύριο. Πιο βασική συζήτηση στην ημερήσια διάταξη τη τελευταία συνεδριάσεω τη ΛΥΜΠΕ πριν τι θερινέ διακοπέ είναι η παρουσία εδώ που μα τιμά των εκπροσώπων τη Λουθουανική ε, Προεδρία. Του καλωσορίζουμε θερμά. Θερμά. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Μπαρνατόνης, Υπουργό Δικαιοσύνης της Λιθουανίας και τον κύριο Μπαρακάουσκας, Υπουργό Εσωτερικών της Λιθουανίας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε έτοιμοι να παρουσιάσετε ε, τις προτεραιότητες της αναλασσόμενης Προεδρίας, της Λιθουανικής Προεδρίας τώρα. Ο κύριος Μπαρακάουσκας έλεγε ότι ξεπερνά κάποια προβλήματα υγείας και έκανε προσπάθεια για να μην χάσει την ευκαιρία και το καθήκον να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της θητείας της Λιθουανικής που αναλαμβάνει την ε, προεδρία μάλλον του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Πολύ σημαντική καμπή αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικές ε, διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται. Πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το τέλος της ηττία και τι ευρωεκλογέ του 2014. Πολλά σχετικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, προστασία των δεδομένων, ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας, νέος κανονισμός της Ευρωπόλ. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συζητηθούν και θα αναφερθούν από τους ομιλητές μας. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, ουσιαστικό είναι ο χρόνος όμως, διότι πλησιάζουμε στην τελική ευθεία της θητείας και όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν ολοκληρώσουμε τα καθήκοντά μας, κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας μικρές πιθανότητες θα υπάρξουν να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά μέχρι το τέλος της θητείας μας. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που ήρθατε. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με τη Λιθουανική Προεδρία και δίνω το λόγο και στους δύο υπουργούς. Πρώτα ο κ. Μπερνατώνης έχει το λόγο σαν Υπουργός Δικαιοσύνης. Α, ο κ. Μπαρακάουσκας πρώτος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Και μετά ο κ. Μπερνατώνης. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πολλούς από εσά εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών και όλους τους παρόντες. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που είμαι εδώ μπροστά σας, προσωπών το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες και τα σχέδια της Λιθουανικής Προεδρίας στον τομέα εσωτερικών, καθώς και τις βασικές ε, προκλήσεις που μας περιμένουν κατά τη διάρκεια του επομένου εξαμήνου. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η πρώτη φορά από όταν προσχώρησε η Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 που αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι μεγάλη τιμή και είναι ιδανική ευκαιρία για να, και ευθύνη βέβαια να εκπροσωπήσουμε τη Λιθουανία. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή για την χώρα μας η αντίληψη των ευθυνών που έχουμε στους ώμους μας Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή και καταβάλαμε πολλές προσπάθειες για να προετοιμάσουμε αυτή, αυτό το σημαντικό γεγονός. Πιστεύω ότι είμαστε ε, απόλυτα προετοιμασμένοι για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τα μέλη του Κοινοβουλίου. Συνέπεια και συνέχεια των εργασιών ειλικρινής διαπραγματεύσεις και συμπερίληψη όλων των σχετικών φορέων σε αυτή τη διαδικασία. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές για την Προεδρία μας, προσπαθώντας να πετύχουμε τον πρωταρχικό μας στόχο να οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη, αναπτυσσόμενη και ανοιχτή Ευρώπη. Θα ήθελα να σημειώσω ότι θα συνεχίσουμε την εφαρμογή του 18 μηνου προγράμματος ε, του τρίο της Προεδρίας και να εργαστούμε προς την επίτευξη των βασικών στόχων που έχουν τεθεί. Ενεργά θα επιδιώξουμε την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις, δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους που είναι οι πιο επίγοντες σε αυτή τη φάση. Δηλαδή θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί στην παρούσα οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση και τις προκλήσεις. Το έργο του Συμβουλίου στον τομέα των εσωτερικών αναμφισβήτητα θα ευθυγραμμιστεί προς την επίτευξη των στόχων και με βάση τις αρχές που προανέφερα. Θα ήθελα να τονίσω ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας η στενή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έγινε ακόμα πιο σημαντική για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνη και των εσωτερικών. Στη δυνατότητα να συνεργαστούμε και το τονίζω αυτό, συνεργαζόμενοι λοιπόν επιτυχώς, πάνω σε αυτή τη συνεργασία βασίζεται η ασφάλεια και ευμάρεια πάνω από 500 εκατομμύρια, για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και όλους τους επισκέπτες της Ένωσης, καθώς και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το χρωστάμε στους πολίτες της Ευρώπης να πετύχουμε τα αποτελέσματα που σωστά περιμένουν από μας. Τώρα που ο κύκλο ο νομοθετικό πλησιάζει προ το τέλο του, ο παρόν, και η Λιθουανία θα είναι η τελευταία προεδρία που θα υπηρετήσει το πλήρε εξάμεινο πριν ε, τις επικείμενες ευρωεκλογέ, βλέπω ότι υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει σε όσο το δυνατόν περισσότερε νομοθετικέ προτάσει. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε ειλικρινεί εκπρόσωποι του Συμβουλίου και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξέβρεση λύσεων που είναι αποτελεσματικές και εξίσου αποδεκτές και στις δύο πλευρές. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό για ενεργό και επικοδομητική συνεργασία. Ήδη το κατανόησα αυτό από πρώτερες επισκέψεις μου στις Βρυξέλλες και εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είμαστε εδώ όχι απλώς για να σας μιλήσουμε για τις προτεραιότητές μας, αλλά επίσης να ακούσουμε και από εσά ποιε είναι οι δικές σας προτεραιότητες, ποιε είναι οι δικές σας ανησυχίες. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον από την αρχή και να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή βάση για πραγματική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα είναι το Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και πρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα ήθελα να αναφερθώ στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει όσον αφορά τον τομέα των εσωτερικών και να περιγράψω διάφορα οριζοντίου φύσεως ζητήματα και ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα εσωτερικών και ασφαλείας και δικαιοσύνης ένα από τα βασικά ζητήματα είναι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ομαλή συνέχιση της οικονομικής ενισχύσεως για τα διάφορα μέσα που εφαρμόζουν τις στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα των εσωτερικών και πρέπει να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία όσον αφορά όλους τους δημοσιονομικούς κανονισμούς μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους το αργότερο. Από την πλευρά μου μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεργαστούμε μαζί σας ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τα, όσον αφορά τα εκρεμή ζητήματα και θα προσπαθήσουμε να θετηθούν όλες οι απαιτούμενε νομοθετικές πράξεις για την ομαλή χρηματοδότηση των θεμάτων εσωτερικών στην νέα συνομική προπτική. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ένα πολύ ευρύ πλαίσιο για τη συνεχή ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης που είναι ένας από τους βασικούς κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω εφαρμογή αυτού του προγράμματος και το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από αυτό το πρόγραμμα θα είναι βασικός στόχος για τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το 2014 είναι το τελευταίο έτος για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αυτό όχι μόνο μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε την σωστή επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος πιο ενεργά, αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ενδεχόμενους μελλοντικούς στόχους για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Μετά από τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα ξεκινήσουμε πολιτικές διαβουλεύσεις όσον αφορά τις ενδεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών μέσω αξιολογήσεως των επιτευγμάτων και στατηγικών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη για το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που θα γίνει στο Βίλνιους στις 18 και 19 Ιουλίου και πραγματικά, πραγματικά ελπίζω να σας δω εκεί ε, και εσάς κύριε Πρόεδρε, κύριε Αγγιλάρ. Το υποσχεθήκατε και θα χαρώ πολύ να ακούσω τη διαβεβαίωσή σας ότι πράγματι θα είστε παρόν σε αυτή την συνάντηση. Τώρα όσον αφορά τα θέματα εσωτερικών, στον τομέα των εσωτερικών, η Προεδρία μας θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα προστασίας των εξωτερικών συνόρων, της νόμιμης μετανάστευσης, της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα στις βασικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητές μας σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, καθώς και στα σχέδια και τους στόχους της Προεδρίας μας που σχετίζονται με αυτούς τους στόχους. Λοιπόν, ένας από τους βασικούς στόχους, προτεραιότητες για τη Λιθουανική Προεδρία θα είναι η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στο στόχο να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανοιχτή, αξιόπιστη και ασφαλή. Η δημιουργία τρόπου διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων δεν είναι μόνο προς όφελος των χωρών του χώρου Σέγγεν, αλλά για όλες τις χώρες είναι υποφελές που δεν έχουν εσωτερικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή που θα σταματήσουν τους ελέγχους στο μέλλον. Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλημάτων, όπως είναι η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση και η διεθνής, ε, το διεθνές έγκλημα και ενισχύεται η γενική εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να ε, αφιερώσουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια για να συζητήσουμε το πακέτο το νομοθετικό για τα ΕΦΗ e σύνορα. Οι πρώτε θέσει των κρατών μελών στο Συμβούλιο έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν σημαντικέ ανησυχίε όσον αφορά την ενδεχόμενη ισορροπία μεταξύ κόστου και όφελου των προτινόμενων συστημάτων κυρίως όσον αφορά την, το πρόγραμμα για την καταχώρηση των ταξιδιωτών. Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες. Έχοντας αυτό υπόψη, σχεδιάσαμε εντατικό πρόγραμμα για τη συζήτηση του πακέτου για τα ευφύη σύνορα στα διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο. Άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η πρόταση κανονισμού που κατατίζει κανόνες για την εποπτεία και έλεγχο των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε πλήρω τη σημασία που έχει αυτή η νομοθεσία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα εφαρμοστεί πλήρω το ταχύτερο δυνατόν. Να πω και μερικά λόγια όσον αφορά το χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τα συγχαρητήριά μου προς την Ιρλανδική Προεδρία και προς όλους εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρήκατε μια λύση για τη διακυβέρνηση του νομοθετικού πακέτου για το χώρο Σέγγεν που ελπίζουμε θα μα επιτρέψει να ξαναρχίσουμε τι παγωμένε διαπραγματεύσει που αφορούν άλλες σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Τώρα, μετανάστευση, για να γίνει πιο ανοιχτή η Ευρώπη, είναι κρισίμου σημασία να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματική πολιτική για τη μετανάστευση. Είμαι πεπισμένο ότι ειλικρινεί ε, και αξιόπιστοι πολίτε από τρίτες χώρε που έρχονται να εργαστούν και να μελετήσουν, να εργαστούν και να μελετήσουν, επαναλαμβάνω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να σπουδάσουν, θα πρέπει να, έχουν, να διευκολυνθούν όσον αφορά την άφηξή του και το ταξίδι του αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής θα συμβάλλει επίσης στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βοηθήσει να καλύψει τις ειδικέ ανάγκες της αγοράς εργασίας και έτσι θα ωφεληθεί η ανάπτυξη της Ευρώπης. Γι' αυτό θέσπιση νομοθεσία στον τομέα της νόμης μετανάστευσης θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Προεδρία μας. Χαιρόμεθα διότι κατά τη διάρκεια τη Ιρλανδική Προεδρία οι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο όσον αφορά του οδηγία του εποχικού εργαζομένου ε, πρακτικά ολοκληρώθηκαν και πετέχθη σημαντική πρόοδο προ μια συμφωνία όσον αφορά την οδηγία για ε, μεταφορέ προσωπικού ε, μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ εταιριών. Έκανε έξοχη δουλειά ο εισηγητή ο κ. Γιακολίνο και ο κ. Μωράε και αυτή είναι μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει και ελπίζω ότι με ενεργό συνεργασία μπορούμε να βρούμε λύσεις όσον αφορά τις εναπομένουσες λεπτομέρειες και αυτή η οδηγία, αυτές οι οδηγίες θα εκτεθούν τάχιστα. Προσβλέπουμε επίσης συνεργασία με την κυρία Βίξτρομ εξετάζοντας ε, την οδηγία για τους φοιτητές και τους ερευνητές και να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο σε αυτό το τομέα. Βεβαίως θα δώσουμε τη δέουσα προσοχή και στα θέματα της παράνομης μετανάστευσης. Σε αυτό το τομέα θα ήθελα να υπογραμμίσω την επικαιροποίηση του σχέδιου δράσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τίτλο «Δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τις μεταναστευτικές πιέσεις, στρατηγική απάντηση». Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, το αυξανόμενο άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτεί επίσης εντατικοποιημένες δράσεις που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών μας και των φιλοξενουμένων της Ενώσεως. Μόνο εγγυόμενοι την ασφάλεια μπορούμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συνεπώς, πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της επιβολής του νόμου και συνεργασία στον τομέα και την ενίσχυση της καταπολέμησης κατά σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας θα είναι ανάμεσα στις ύψιστες προτεραιότητες τη Προεδρίας μα. Να πω και κάποια θέματα για τον κανονισμό περί Ευρωπόλ. Ιδιαίτερη, μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με αυτό το θέμα είναι η πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη συνεργασία των δυνάμεων της τάξης και την κατάρτιση. Είναι το πρώτο σημαντικό νομοθετικό χαρτοφυλάκιο μετά τη συνθήκη τη Αβώνας επηρεάζει την συνεργασία των δυνάμεων επιβολή του νόμου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που προσπαθούν να καταπολεμήσουν το σοβαρό και οργανωμένο διεθνέ έγκλημα καθώ και την αντιμετώπιση προβλημάτων εσωτερική ασφαλείας εν γέννη. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό έχει πολύ σοβαρή και υπεύθυνη στάση όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία και το Συμβούλιο ξεκίνησε εντατικέ εργασίε για να εξετάσει και να συζητήσει την πρόταση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Οι συζητήσει στο τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι κατά τη προτάσεω συγχώνευση τη ΕΠΟΛ και με την Ευρωπόλ. Και θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία μα θα επιδιώξει να πετύχει σημαντική πρόοδο μέσω εντατική εξέταση τη προτάσεω στο Συμβούλιο σε επίπεδο πολιτικό αλλά και επίπεδο επαϊόντων. Άλλο νομοθετικό χαρτοφυλάκιο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλά κράτη-μέλη είναι το θέμα ε, των, για τα στοιχεία επιβατών PNR. Ο μηχανισμός μεταφοράς των στοιχείων ήδη λειτουργεί μέσω διμερών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τη ΣΥΠΑ, με την Αυστραλία και τον Καναδά. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, είναι ζωτική σημασίας να έχουμε εσωτερική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα PNR τα στοιχεία επιβατών με λόγια. Υπάρχουν ε, μεγάλε προσδοκίε για περαιτέρω διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το ευαίσθητο αυτό θέμα και προσωπικά σα ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να μας βοηθήσετε στη δουλειά αυτή. Μέσω αμοιβαία επικοδομητική συζήτηση θα μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Τώρα η τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επικίνδυνο, κατεπήγον, μεγάλη απειλή για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για την ασφάλεια των πολιτών της. Γι' αυτό η Προεδρία μας θα φωσιώσει, θα δώσει μάλλον ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δίνοντας έμφαση σε ορισμένες πτυχές της πρόληψης ε, του βίου εξτρεμισμού, ε, ριζοσπαστικής προσέγγισης, ε, ε, Στρατολόγηση τρομοκρατών και χρηματοδότησης των τρομοκρατών και το ευαίσθητο θέμα των αποκαλούμενων ξένων μαχητών, αλλοδαπών μαχητών. Υπάρχουν πολλά νέα πράγματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να πω ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι περιπλοκότατη πρόκληση που όλο και περιπλέκεται, άρα θα εργαστούμε άοκνα σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της κυβερνοασφαλείας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που θα λάβει η χώρα ε, στο Βίλνιους και σε, διάφορες άλλες, σε διάφορα άλλα βήματα σχετικά θα ήθελα να τονίσω ότι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι μια πρόκληση παγκοσμίου φύσεως. Γι' αυτό θα καταβάλουμε προσπάθειες για να βρούμε λύσεις όχι μόνο εσωτερικώς αλλά και μέσω διεθνούς συνεργασίας μαζί με τους στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να πω και δύο λόγια για την εξωτερική πολιτική Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στον τομέα τη δικαιοσύνη και εσωτερικών, ενισχύοντα τομεακή συνεργασία με τρίτε χώρε και συνεχίζοντας συνεχί, το πολιτικό διάλογο με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε να ετοιμάσουμε παραδοσιακή υπουργική συνεδρίαση των Υπουργών εσωτερικών και Δικαιοσύνης με συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα με τι χώρε τη ανατολική ε, γειτονία. Θέλουμε να επεκτείνουμε τον τομέα τη εσωτερική μα ασφαλεία πέρα από τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, οικοδομώντα αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Υπό το φως αυτού σχεδιάζουμε να διεξαχθεί το πρώτο Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Ενώσεω με τις χώρες της Ανατολικής ε, Συνεργασίας σε διπουργικό επίπεδο για να συζητήσουμε τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Και τώρα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα να πω όσο δυνατόν περισσότερα, ώστε να μην υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις που θα μου θέσετε. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφό μου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τη Δημοκρατία τη Λιθουανία, τον Γιώζα Μπερνατόνη, ο οποίο θα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη Προεδρία μα στον τομέα τη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε για την ε, παρουσίασή σα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Βίλνιους ε, και θα εκπροσωπήσω εκεί την ε, Επιτροπή Λίμπε. Θα δώσουμε τώρα στον κύριο Μπερνατόνη τώρα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μας μιλήσει αυτός για το πρόγραμμα της ε, Λιθωνικής Προεδρίας. Επιτρέψτε μου, ε, όπως και ο κ. Μπαρακάουσκας, να εκφράσω και εγώ την επιθυμία μας και την προθυμία μας να συνεργαστούμε μαζί σας το επόμενο εξάμεινο. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Άρα θα ήταν καλό να εξασφαλίσουμε από την αρχή μια καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας στην προετοιμασία της Προεδρίας μας, ιδιαίτερα για την πολύ χρήσιμη συνεδρίαση του ε, Μαρτίου, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Αγγιλάρ, ε, μας ε, βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Αναμένουμε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και όλο το εξάμεινο της Προεδρίας μας. Είναι σημαντικό να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, ε, ευρωπαϊκή αγορά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και γενικότερα την οικονομία μας. Ε, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την νομική βάση για την προστασία των δεδομένων. Για... Θα διοργανώσουμε μάλλον μέσα το Δεκεμβρίου στο Βίλνιους και μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε το τι έχει, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών και να χαράξουμε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον σε αυτό τον τομέα. Θα εστιαστούμε στα νομοθετικά μέτρα για θέματα δικαιοσύνης έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ε, και την περίοδο την οποία διανύουμε. Το πακέτο προστασίας των δεδομένων από την άλλη μεριά είναι ένα πολύ περίπλοκο ε, πακέτο. Έχει ως ε, στόχο να εξορροπήσει τα συμφέροντα των, του ατόμου και ταυτόχρονα να, με την οικονομική ανάπτυξη. Η Προεδρία θα συνεχίσει την εξέταση του κανονισμού και της οδηγίας ως πακέτο. Ε, ελπίζουμε ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον κανονισμό. Ενώ σε ό,τι την οδηγία. Επίσης θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, υπάρχουν εκεί διατάξεις ειδικά, ειδικά για την εφαρμογή του νόμου. Για την μεταρρύθμιση προστασία δεδομένων μπορώ να πω ότι ε, θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι περίπλοκη, θα επηρεάσει πολλούς τομείς, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν Δεν θα πρέπει να κάνουμε προχειρότητες για να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Το χρονοδιάγραμμα για το πακέτο προστασίας δεδομένων είναι πολύ ε, φιλόδοξο. Σας διαβεβαιώνω ότι θα αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθειες για να προχωρήσουμε αυτό το πακέτο. Με τον κύριο Άλμπρεχτ και τον κύριο Δρούτσα έχουμε ήδη επαφές που είναι εισηγητές. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω του ποινικού δικαίου έχουμε ήδη πρωτοβουλίες ε, οι οποίες σύντομα θα ξεκινήσουν. Να αρχίσω από την οδηγία για την καταπολέμηση ε, της απάτης έναντι των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η πρόταση αυτή έχει ως σκοπό να ε, εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Το Συμβούλιο θα θυμάστε ότι είχε καταλήξει μια κοινή προσέγγιση για το σχέδιο οδηγία. Τα κράτη-μέλη είχαν εκφράσει επιφυλάξει για ορισμένα πράγματα όπως η νομική βάση της πρότασης, ο ορισμός της ε, απάτης, ε, ο χρόνος παραγραφής και κάποια άλλα θέματα. Ε, για όλα αυτά το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αναμένουμε την εκθέσει των ε, αρμόδιων επιτροπών και ήδη είμαστε έτοιμοι για ε, άτυπες επαφές με τον κύριο Αγγιλάρ που είναι ο, ο εισηγητής. Ε, αυτό το θέμα πάει χέρι-χέρι με την μελλοντική πρόταση Κομισιόν για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Δημιουργήθηκε από την συνθήκη της μια ειδική νομική βάση γι' αυτό. Το θέμα το συζητούμε όλη την τελευταία δεκαετία. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να γίνουν επικοδομητικά. Το θέμα είναι περίπλοκο. Θα χρειαστεί προσπάθεια και χρόνος και από τα κρατημέλη και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο θα συμπεριλάβανε επίσης και ε, ένα κείμενο για την ε, μεταρρύθμιση της Eurojust, της δομής της Eurojust. Η Προεδρία έχει στόχο οι συζητήσεις να γίνουν παράλληλα για τα δύο θέματα. Οι πρώτες συζητήσεις θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Η οδηγία για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων εναντί παραχάραξης μέσω του ποινικού δικαίου έχει στο σκοπό να ενισχύσει την αξιόπιστη Ευρώπη. Η οδηγία αυτή θα αποτελέσει για μας προτεραιότητα. Το μέσο αυτό θα εξασφαλίσει σταθερότητα και ε, προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της παραχάραξης. Η Προεδρία αναμένει να γίνει στο Συμβούλιο μια επικοδομητική συζήτηση αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο. Αναμένουμε και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και τη ηγέτης τη Κυρία Μάκινταρ. Η Προεδρία θα εργαστεί επίσης και, και επί οδηγίας για την ε, δίμευση και, ε, κα, και ε, ανάκτηση προϊόντων εγκλήματο μέχρι το τέλος του χρόνου. Η υιοθέτηση ευρωπαϊκών ελάχιστων κανόνων για την κατάσχεση και τη δίμευση ε, τέτοιων προϊόντων εγκλήματος είναι σημαντικό βήμα για να ε, αποφύγουμε ε, τις εγκληματικές δράσεις. Κυρία Μάκοβε είναι η συγκητρία. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν σε μια συνένεση αποδεκτή από όλου. Με πολύ ικανοποίηση σημειώνουμε ότι η πρώτο της Ιρλανδική Προεδρία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας ε, ήταν σημαντική. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είχε ως ε, στόχο ένα ομοιόμορφο σύστημα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων για όλες τις ποινικέ υποθέσεις. Ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας θα αποτελέσει ένα ε, χρήσιμο εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα είμαστε σε επαφή με τον κύριο Μέλο, τον εισηγητή και με όλο το κοινοβούλιο, προκειμένου να καταλήξουμε στη συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Παρόλες τις προκλήσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι έτοιμη. Ε, μία από τι οριζόντιε προτεραιότητε τη Προεδρία, όπω είπε ο κ. Μπαρασκάουσκα, ε, είναι ε, η ενίσχυση τη συνεργασία με τις ανατολικέ γειτονικέ χώρε στον τομέα τη δικαιοσύνη. Από την πρώτη μέρα τη Προεδρία μα ήταν σαφέ ότι θα αντιμετωπίσουμε και θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα τη Προεδρία, που έχουν γίνει όμω πολύ επίκαιρα και πιεστικά. Για παράδειγμα, οι πληροφορίε για το πρόγραμμα παρακολούθησης εκ μέρου τη Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλεία των ΗΠΑ. Αυτό το θέμα γύρει σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ο διάλογος με τους Αμερικανού εταίρου μας ξεκίνησε χτε στην Ουάσιγκτον και η Κορεπέρα αύριο θα συζητήσει το ζήτημα ξανά. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες της ε, Προεδρίας της τόν τομέα της ε, δικαιοσύνης. Δεδομένου ότι ο νομοθετικός κύκλος του Ευρωκοινοβουλίου φτάνει στο τέλος του, ε, θα πρέπει να πιέσουμε προς μια επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή σε διάφορα ντοσιέ, σε διάφορους φακέλους σε συνεργασία, αν συνεργαστούμε μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της Προεδρίας. Με χαρά θα καλωσορίσουμε μέλη της Επιτροπής σας την επόμενη εβδομάδα στο Βίλνιους, στο άτυπο ε, Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ε, μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας αν υπάρχουν, να ακούσω τα σχόλιά σας κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο σας, κύριε Μπαρακάουσκας και κύριε Μπερνατώνης. Σίγουρα από τις ε, λεπτομέρειες που μόλις μας παρουσιάσατε έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη διαφορά σε αυτή την ε, νομοθετική περίοδο. αυτή η τελική ευθεία που είναι η δική σας προεδρία μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη να σας υπενθυμίσω μόνο ότι το πρόγραμμά μας προέβλεπε να διαρκέσει η συζήτηση μέχρι τις 4 και 4. Μετά έχουμε καλέσει την ε, Ιταλίδα Υπουργό Ένταξης. Φυσικά μπορούμε να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα, όμως θα σας παρακαλούσα να είστε όσο το δυνατόν συντομότεροι. Έχω τον κατάλογο των ομιλητών. Σας προτείνω να εχετε δυο δύο-τρία λεπτά στη διάθεσή σας ο καθένας. Η κυρία Ματιέ αρχίζει ως ε, συντονίστρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργή. Λοιπόν, όσο μας αφορά, Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμεθα εδώ, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, όπως είπε και ο Πρόεδρος, φτάνετε σε μια στιγμή της θητείας κρισίμου σημασίας. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε κάποια χαρτοφυλάκια σημαντικότατα. Euh, Τον επόμενο χρόνο τα χαρτοφυλάκια θα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, θα έχουν σταματήσει. Για μας κάποια θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά Κάποια ήδη ολοκληρώθηκαν. Αναφερθήκατε κύριε Υπουργέ για το Σέγγεν. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτά που έγιναν στον αφορά του Σέγγεν. Υπάρχει καλύτερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, περισσότερη ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μετά ελεύθερη μετακίνηση που θεωρείται και εκτιμένη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θέλαμε και αυτό πετύχαμε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιτευχθή σας συμφωνία. Αναφερθήκατε στη μετανάστευση, μετανάστευση οικονομικού χαρακτήρα. Θέλουμε με την έκθεση που έχουμε επιτάπητος και ελπίζουμε να αποπερατωθεί κατά τη διάρκεια της Λιθανικής Προεδρίας. Θέλουμε να έχουμε αποτελεσματική μετανάστευση που να είναι συντονισμένη για τα άτομα που έρχονται να εργαστούν, να σπουδάσουν και θέλουμε τα δύο χαρτοφυλάκια τα αντίστοιχα προς το τέλος της αυτά που πρέπει να συζητηθούν να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Αναφερθήκατε στι ΕΠΟΛ και την Ευρωπόλ. Είχαμε την παρουσίαση της εκθέσεως του εισηγητού της Ευρωπόλ, σήμερα το πρωί το συζητήσαμε. Οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε είμαστε κατά τη συγχώνευση ΕΠΟΛ-Ευρωπόλ. Από τη μια, διότι δεν θα υπάρχει προστιθέμενη αξία για να γίνει αυτή η συγχώνευση. Και μετά από την άλλη, διότι θέλουμε τη διόνυση, τη συνέχιση τη κατάρτιση τη αστυνομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάποια κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη μάλλον, επιθυμούν η αστυνομία να μπορεί να συνεχίσει την κατάρτισή της μέσω αυτής της, αυτού του ωραίου μικρού οργανισμού της ΕΠΟΛ οπότε αυτό το συζητήσαμε λίγο σήμερα το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να το πούμε κάποια θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά για μας τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων οδηγία και κανονισμός το θέμα της Ευρωπόλ που προανέφερα και βέβαια το PNR, τα στοιχεία επιβατών που θέλουμε και αυτό να προχωρήσει και θέλουμε προφανώς να γίνουν πολλές προσπάθειε και μας απασχολεί εμά το ΕΛΚ. Το θέμα της κατάσχεσης των εσόδων από το έγκλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Το θέμα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας και αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα για την ε, ριζοσπαστική τοποθέτηση των νέων ε, που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για μας να καταλήγουν σε ακραίες θέσεις οι νέοι με άλλα λόγια έκανε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς το ίδιο για την ένταξη των Ρωμά, των πληθυσμών Ρωμά. Αυτό είναι και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, το προσέχουμε, αυτή η ένταξη των πληθυσμών των Ρωμά. Θέλουμε να το λύσουμε, συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο Γιαρόκα. Αν μπορούσατε κι εσείς να φροντίσετε τόσο αυτό να αποκτήσει κάποια ουσία και εύρος, θα σας είμαι θα ευγνώμονες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μποσκούρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω. Η μία έχει να κάνει με την ε, απάτη, την οικονομική απάτη. Μας είπατε ότι στις προτεραιότητές σας ε, θα είναι ορισμένες οδηγίες σχετικά με την απάτη, όμως ε, λείπει, λείπουν και ρυθμίσεις σχετικά με την κατάχρηση στον χώρο της αγοράς, που είναι εξίσου σημαντική. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης κάποιων κανονισμών πάνω σε αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω η ανάκτηση εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς ε, οραματίζεστε εσείς τον τριμερή διάλογο για αυτό το θέμα, διότι το Κοινοβούλιο έχει λίγο πολύ εννέα θέση, αναρωτιέμαι όμως ποια είναι η θέση της Ελληνικής Προεδρίας και τι προτίθεται να κάνει και ποια είναι η φιλοδοξία σας. Φιλοδοξείτε όπω και η Ιρλανδική Προεδρία στο τέλος της θητεία σας να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για την οδηγία αυτή. Μετά, η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει με την, τον πόλεμο κατά των διακρίσεων. Υπάρχει σχετική οδηγία, αλλά τι γίνεται με την οδηγία αυτή. Υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχει κάποια φιλοδοξία για να προχωρήσει το θέμα, διότι τα τελευταία πέντε χρόνια γίνονται διαβουλεύσεις και πιστεύω ότι για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Κύρια Βέμπερ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, κύριους Υπουργούς για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Λιθουανικής Προεδρίας. Είναι αρκετά φιλόδοξο το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε και σας εύχομαι καλή τύχη. Εάν τα καταφέρετε, τότε πραγματικά θα έχετε ενεργήσει προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Τουλάχιστον για κάποιες από τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον καθέναν από εσάς και για τους δυο σας. Καταρχάς να πω ότι καλωσορίζω το ότι αναφέρατε ότι η προστασία δεδομένων θα ε, συζητηθεί ως ε, ένα ενιαίο πακέτο, διότι και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή να ε, ε, τύχει επεξεργασία ταυτόχρονα με τον κανονισμό. Επίσης, όπως και ο συνάδελφός μου, έχω και εγώ την, μια παρόμοια ερώτηση. Τι γίνεται με την οδηγία κατά των διακρίσεων καταπολέμηση των διακρίσεων είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για την ε, δική μου πολιτική ομάδα. Και όσον αφορά την ε, ομοφοβική νομοθεσία, τουλάχιστον έτσι θεωρούταν στην ε, Λιθουανία για, τις, για τα φεστιβάλ των ομοφιλοφίλων, θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια των ε, Θα ήθελα να πω λοιπόν να ρωτήσω τι γίνεται εκεί τώρα. Όσον αφορά τη συζήτηση με τους Αμερικανούς εταίρους μας, να σας πω ότι το θέμα δεν είναι μόνο το PRISM και το, αυτό το πρόγραμμα, αλλά το τι έχουν κάνει και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης, ποιες είναι οι δικές τους ευθύνες στο θέμα αυτό και αναρωτιέμαι εάν στην ομάδα εργασίας θα αντιπροσωπεύεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, προς τον ε, κύριο Μπαρακάουσκας, θα ήθελα να πω ότι καταρχάς πρέπει να παραδεχτώ ότι η δική μου ομάδα δεν θεωρεί ως προτεραιότητα τα δεδομένα των επιβατών, τα PNR. Ήδη έχουμε πει ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί το πακέτο με την προστασία των δεδομένων και τη σχετική οδηγία πριν από τα δεδομένα των επιβατών. Όμως, θα με ενδιέφερε ε, να μάθω τι γίνεται σχετικά με τα δεδομένα των επιβατών και τη Ρωσία. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πληροφορία για το θέμα αυτό και μέχρι τώρα ήταν δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να μάθουμε οτιδήποτε και να τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία για τον ε, νέο κανονισμό για τα PNR που έχει προωθήσει η Ρωσία. Και τέλος, μία ερώτηση για την ε, προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο του Σέγγεν. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε όλοι ότι οι δύο αυτές χώρες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, εσείς προσωπικά ή η Λιθουανική Προεδρία γενικότερα έχετε κάποια στρατηγική για να πείσετε τα πιο διστακτικά κράτη-μέλη να δεχτούν τις δύο χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, κυρία Φλότχα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Υπουργή. Καλώς ήρθατε. Είσαστε προφανώς ευτυχείς να είστε μαζί μας και είναι κοινή αυτή η χαρά. Η συνεργασία είναι η αφετηρία της υλοποίηση που, των σχεδίων που είναι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών φτάσατε το ξέσπασε η υπόθεση Σνόντεν και η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στις σχέσεις που ε, έχουμε με τη ΣΥΠΑ είναι ένα θέμα που αφισβητείται και θα έλεγα αφισβητείται πολύ είναι πολύ πιο δύσκολο να, να Είναι πιο εύκολο να περάσει παράνομο ε, αεροπλάνο της CIA ελεύθερα από τον ενέργειο χώρο από ότι είναι να περάσει το προεδρικό αεροπλάνο. Λοιπόν, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε δικαιολογία την καταπολή τη τρομοκρατία. Μία από τι χώρε, από τι σπάνιε χώρε, τι ευρωπαϊκέ, που πήρατε το θέμα τη παράνομη ε, μεταφορά κατά ε, υπόπτων από τη CIA στα σοβαρά. Έχετε ενεργήσει δύο έρευνε όσον αφορά τι παράνομες αυτέ επιδόσει και είστε οι χώρες που καλύτερα θα μπορεί να δώσει μια πρόθεση στο Συμβούλιο ε, ούτω ώστε να επιτευχθεί αυτό που ζήτησε με πλειοψηφία τον περασμένο Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο και που θα συζητήσουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο, δηλαδή κάτι που αφορά τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την αναγνώριση συμμετοχή των κρατών μελών, όσον αφορά το πρόγραμμα της CIA, το παράνομο, των παρανόμων επιδόσεων. Να περιμένω να ακούσει ο Υπουργό Εσωτερικών, εδώ είμαι κύριε Υπουργέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ε, Θα τα πω γρήγορα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στο, από πλευρά Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου και από πλευρά του Συμβουλίου Υπουργών. Ποιε πρωτοβουλίε θα αναλάβετε, ούτω ώστε όπω είχε ζητήσει με μεγάλη πλειοψηφία το Σεπτέμβριο τον περασμένο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα μπορέσει να γνωστοποιήσει ποια είναι η συμμετοχή των κρατών μελών όσον αφορά το παράνομο πρόγραμμα των επιδόσεων τη CIA το 2001 και μετά και να βοηθήσετε τι χώρε όπω η δική σα που κάνουν έρευνε και ήσασταν πάντα ανοιχτοί να ξανανοίξουν οι έρευνε. Πρώτη έρευνα περιορίστηκε στο στόχο ε, στην κατάχρηση εξουσία και για τι εξαφανίσει και τη βασανιστήρια δεν έκανε έρευνε, είναι όρια. Νέα στοιχεία μέσω των στοιχείων του Ευρωκοντρόλ υπάρχουν. Έχετε τα στοιχεία σα, τα διαβίβασα, διαβιβάστηκαν στου εισαγγελεί και στι αρχέ. Έχετε λοιπόν στα χέρια σα τα μέσα να γίνετε η μεγάλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η οποία θα αποκαταστήσει την τιμή και την εξοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τα θέματα τη εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτε έναντι του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών. Δεύτερον, τι πρωτοβουλίε θέλετε να αναλάβετε, τόσο ώστε να ανταποκριθείτε στην επιστολή που έστειλαν τέσσερι χώρε όσον αφορά έναν εσωτερικό μηχανισμό ευρωπαϊκό, ενδοευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου και αξιολογήσεω τη καταστάσεω όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει τη δουλειά του, θα το θέσουμε στη μερίσια διάταξη τη επόμενη συνεδριάσεω ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία ανακοίνωση όσον αφορά που θα την υποβάλει μετά τι διακοπέ και αναμένεται και το Συμβούλιο θα κάνει. Να θεσπιστεί λοιπόν ένα μηχανισμό αξιολογήσεω για την αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Κίρκοπ έχει το λόγο, που είναι εκπρόσωπο του ECR και εισηγητή για το θέμα αυτό του PNR του Ευρωπαϊκού. Θα είμαι σύντομο. Ζητώ Συγγνώμη, έχουμε μια συνάντηση για τα συνόδευτα παιδιά, του ασυνόδευτου ανηλίκου, κάπου αλλού στο κτίριο, οπότε θα χρειαστεί να φύγω. Θα σα αφήσω το σχόλιο μου. Καταρχήν, να καλωσορίσω θερμά την Προεδρία αυτή και τον κατάλογο με τους στόχους της. Σε ό,τι αφορά το PNR, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Υπουργό, ε, που υποστηρίζει την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν ανησυχίες και για το θέμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει μια σειρά διμερών συμφωνιών να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό χωρίς να το ελέγχουμε. Χρειάζεται να έχουμε ένα κεντρικό έλεγχο ε, μέσω καταρχήν μιας ε, πρότυπης ε, συμφωνίας για τα PNR στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο σχόλιο που έχω να κάνω το εξή. Πιστεύω ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μία από τι προτεραιότητε τη Προεδρία, είναι ένα πράγμα το οποίο πολλοί πολιτικοί και πολλές κυβερνήσεις ε, ε, είχαν προαναγγείλει θεωρητικά, αλλά στην πράξη δεν έκαναν τίποτα δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή πάνε στις τσέπες ε, εγκληματιών ε, εξαιτία του εγκλήματος στην κυβερνοχώρο. Ε, άλλου τύπου εγκλήματα στον 20ο αιώνα τα είχαμε γνωρίσει καλά και μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα έγκλημα του 21ου αιώνα το οποίο μας δυσκολεύει ιδιαίτερα. Αν παραμείνει προτεραιότητα το ζήτημα για εσάς, θα σας υποστηρίξουμε πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία με τα, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα μέλη. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ, για να έχουμε και τις απαντήσεις. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να καλωσορίσω την πρώτη Βαλτική Προεδρία, τους Λουθιανούς Υπουργούς. Το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε είναι πολύ ε, φιλόδοξο, το υποστηρίζω. Ε, ο παράγοντα χρόνος είναι σημαντικός. Παρακαλώ πολύ βοηθήστε μας να προχωρήσουμε θέματα όπως οι εποχιακοί εργαζόμενοι, ε, το θέμα των ερευνητών και των φοιτητών κλπ. Η, η οικονομία της Ευρώπης είναι οικονομία έντασης γνώσης, άρα χρειάζεται να ε, κινητοποιήσουμε τους ερευνητές. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, να το εξής. Και εδώ ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα. Ελπίζω ότι το PNR θα αποσυνδεθεί από το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Και θα ήθελα επίσης ιδιαίτερα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών στο ίντερνετ. Ελπίζω θα καταλάβουμε κάποια στιγμή την διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη δυνατή προστασία δεδομένων και την, ε, τις λειτουργίες μιας μυστικής υπηρεσίας. Είναι κρίμα που Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά αυτή ε, εδώ πέρα. Ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Ελπίζω το πρίσμα ε, να ε, μην κυριαρχεί στη συζήτηση για την προστασία δεδομένων. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία σε ζητήματα, σε ποινικέ υποθέσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Έρευνα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Έντσιου. Να καλωσορίσω τους δύο υπουργούς στην Επιτροπή μας. Καλή επιτυχία το επόμενο εξάμεινο. Είναι συνεισηγητής και σκιοσηγητής για το πακέτο των φιών συνόρων. Να κάνω λοιπόν κάποια σχόλια. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο για την ε, Εσωτερική Ασφάλεια ε, εκεί διαθέτουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τα ευφύ σύνορα. 1,1 δις συγκεκριμένα. Τι θα γίνει με αυτό το πακέτο. Θα καθυστερήσει, θα εφαρμοστεί, πώς το βλέπετε εσείς. Θα καταφέρουμε να το ξεκινήσουμε. Κάποιες πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν με αυτό το πακέτο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λένε ότι τα ωφέλη δεν είναι ανάλογα με, την, με τον προπολογισμό του. Και κάτι άλλο, ένα σχόλιο. Το ανέφερε και η Ρενάτε Βέρβερ. Η είσοδος στην ζώνη Σέγγεν της Ρωμανίας και της Βουλγαρίας ίσως είναι οι δύο χώρες που είναι πιο καλά προετοιμασμένες από τεχνικής πλευράς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ζώνη Σέγγεν. Από το 2011 και μετά όλες οι προεδρίες είχαν θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα αυτό. Ελπίζουμε ότι τελικά θα ολοκληρωθεί η είσοδος της και της Βουλγαρία στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλος αυτή την επιτροπή κανονικά, αλλά παρόλα αυτά θέλω να καλωσορίσω τους υπουργούς μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων που κάνατε. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε κάποια πράγματα. Αυτό δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε στην Επιτροπή ότι ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα. Ένα από τα ζητήματα που ήθελα να αναφέρω είναι η ενεργοποίηση κάποιων μέσων και κάποιων θεσμών όπως το ΣΕΠΟΛ, το θέμα του κανισμού για ΣΕΠΟΛ και Ευρωπολ αναφέρθηκαν και κάποιες κινήσεις και δραστηριότητες του Συμβουλίου. Θα ήθελα λεπτομέρειες όμως. Τι θέλει να κάνει η Λιθουανική Προεδρία όσον αφορά την προστασία των πολιτών, την κυβερνοασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θέλουμε να προστατεύουμε τους πολίτες μας στο βαθμό του δυνατού. Είναι έφτραυστο το περιβάλλον, όμως είναι δύσκολη καιρή. Θεωρείτε ότι η συγχώνευση Ευρωπόλ και ΣΕΠΟΛ είναι κάτι υποφελές ή κάτι αρνητικό. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, άλλο θέμα. Η χώρα μας ε, δέχτηκε επίθεση σε επίπεδο DDoS. Εικάζεται ότι ήταν από χώρα τρίτη. Πώς, πώς φαντάζεστε τη συζήτηση στο Συμβούλιο για να, να βρεθεί ένα σύστημα απάντησης σε αυτές τις απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. λένε κάποιοι ότι οι επιθέσεις DDoS είναι ψηφιακή εκδήλωση απόψεων και όχι έγκλημα. Ε, η δική σας άποψη ποια είναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διαβάζω στο πρόγραμμά σας ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών θέλετε να ανακτηθεί εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και να προστατεύσετε τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν βλέπω όμως λεπτομέρειες. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να το κάνετε. Έπειτα, μας λέτε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ε, για την ολοκλήρωση των ε, διαφορών τυπικότητων και πιστοποιητικών, αλλά πότε. Κύριος Λόπες. Κύριε καλώς Καλωσορίζω και εγώ την πρώτη Βαλτική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς στην Ισπανία ζήσαμε κάποια στιγμή αυτή την σημαντική στιγμή της ιστορίας μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Στον Υπουργό Εσωτερικών θα ήθελα να απευθύνω το εξής ερώτημα. Εξέφρασε την ανησυχία του για το θέμα των εσωτερικών συνόρων. των εξωτερικών συνόρων, συγγνώμη. Ε, έχει σκοπό να εντείνει τη συνεργασία με τρίτε χώρες και δεύτερον σε ό,τι αφορά το PNR καταλήξαμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια η, η, η, οι ε, Αμερικανοί ε, συνδέουν ε, την ασφάλεια των σύνορων τους με την ομοποίηση 11 ε, εκατομμυρίων λαθρέων μεταναστών εκεί. Ποια είναι η άποψή σας ε, σε σχέση με αυτό το θέμα και σε σχέση με τη δική μας διαχείριση εξωτερικών σύνορων. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Αν δεν μιλήσατε για ορισμένες εκκρεμότητε σε ό,τι αφορά τις διαδικαστικές εγγύησεις για το θέμα για παράδειγμα της ε, ε, δωρεάν συνδρομής ε, και για το τεκμήριο Ε, Γνωρίζετε ότι οι συνθήκες κράτησης δεν είναι σημαντικές μόνο στην Ευρώπη. Είναι και για όλους. Τι γίνεται με τους ετούντες άσυλο που κρατούνται κοντά στα σύνορα ή στα σύνορα. Ποια είναι οι προθέσεις σας δεν μιλούμε μόνο για τις συνθήκες κράτησης των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να μιλάμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στα κέντρα κράτηση στα σύνορα. Παρα... Παρακαλώ. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Κύριε Μπρόνς, πρώτο κύριος Μπάτεν και έπειτα ο κύριος Μπρόνς. Κύριε Μπάτεν, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Θα είμαι σύντομο. Ορισμένε ερωτήσει που ήθελα να κάνω ήδη τι ανέφεραν οι συνάδελφοι. Καταρχά, ποια είναι η άποψη τη Λιθουανική Προεδρία για τη συγχώνευση Ευρωπόλ και ΣΥΠΟΛ. Είστε υπέρ κατά αυτή τη συγχώνευση. Μετά, όσον αφορά τα έξυπνα σύνορα και το πακέτο αυτό, πιστεύετε ότι οι αρχές επιβολής ενόμου εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα εισόδου και εξόδου όπως προβλέπεται από το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα και τι πιστεύετε για το πακέτο αυτό. Τρία. Σέγγεν. Ποια είναι η άποψή σας για τη διεύρυνση της περιοχής του Σέγγεν ε, με τη συμπερίληψη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Σχεδιάζεται κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Έχει η Λιθουανία συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με τις ε, επιπτώσεις του που θα έχει η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ε, στο οργανωμένο έγκλημα. Προβλέπετε κάποιο μηχανισμό για να τους εμποδίσετε αυτές τις δύο χώρες να μπουν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Καταλάβαμε κύριε Μπρόντς, τελευταία ερώτηση καλωσορίζω το γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα στον έλεγχο των εξωτερικών ε, συνόρων και, να, και την ε, αποτροπή της παρανομή ε, μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παρανομ... και της διακίνησης. Ωστόσο δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα το πετύχετε. Δεν υπάρχουν δυνατότητες και χώροι κράτησης αρκετοί για να υποδεχτούν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, ε, καθώς έχουμε πληροφορηθεί από τον Γενικό Διευθυντή της ε, Frontex, όταν κάποιοι μετανάστες ε, δεν καταφέρνουν να πάρουν άσυλο, τους παρέχεται ένα έντυπο, ένα φύλλο χαρτί και μετά τους αφήνουν να φύγουν. Τώρα, όσον Τώρα η διαχείριση της μετανάστευσης έχει σκοπό να ικανοποιήσει την αγορά εργασίας. Υπάρχει όμως μεγάλη ανεργία και δεν υπάρχουν αρκετές ε, θέσεις ε, ώστε να απορροφήσουν αυτούς τους μετανάστες. Υπάρχει μάλιστα ο κίνδυνος ε, στην μετακίνηση εργατικού δυναμικού, η μετακίνηση εργατικού δυναμικού να ταυτιστεί με την παράνομη διακίνηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπρόνς. Μάλιστα, αυτή ήταν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις ε, και οι προσδοκίες από την πρώτη, για την πρώτη Λιθουανική Προεδρία. Πολλά τα ερωτήματα, ξέρω. Σας ε, καλώ τώρα να απαντήσετε όσο δυνατόν πιο συνοπτικά στις ερωτήσεις των ε, μελών. Και σας εύχομαι καλή τύχη. Ο κύριος Μπαρακάουσκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις. Χαίρομαι πολύ που οι ερωτήσεις σας ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αγγίζουν σημαντικά θέματα για όλη την Ευρώπη και αφορούν την, τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Καταρχάς, ε, κυρία Μαλίνοφ, Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Τώρα όσον αφορά το τι θα κάνουμε με την ΕΣΕΠΟΛ, να σας πω ότι στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου στα τέλη Ιουνίου η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν ενέκρινε μια πιθανή συγχώνευση. Ορισμένα κράτη-μέλη πρότειναν να βρεθεί κάποια λύση η οποία θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία και τον δύο οργανισμών, ε, συγχωνεύοντας ίσως μόνο τα διοικητικά τους όργανα. Του χρόνου τις αρχές του Μαρτίου που θα μεταφερθούν τα κεντρικά αυτά στην, ε, στο Βασίλειο ίσως ε, προχωρήσει το θέμα. Η πρόταση αυτή όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστεί από την αρχή. Να σας, διασφαλίσω, να σας διαβεβαιώσω όμως ότι το Συμβούλιο θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την ομαλή λειτουργία και των δύο οργανισμών. Τώρα, κύρια Βέμπερ, από, τη, από τους φιλελεύθερους σας γνωρίζω αρκετά καλά και να πω ότι κάνατε ορισμένες πολύ καλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά το Σέγγεν, μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η προσχώρηση των δύο αυτών χωρών πράγματι είναι κάτι το οποίο ανάμεναμε εδώ και χρόνια και είναι μια ανησυχία για πολλά κράτη-μέλη, διότι άνοιγαν στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Η Λιθουανία ως ε, επίσης πρώην μέλος του Ανατολικού Μπλοκ θα απασχίσει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για έβρεση λύσεις για το θέμα αυτό. Αυτά εν συντομία για το πρώτο ερώτημά σα. τώρα, όσο για το δεύτερο. για τους πολίτες και τα προσωπικά δεδομένα. Νομίζω πως άλλοι τρεις συναδελφοί σας έκαναν την ίδια ερώτηση. πιστεύω ότι εδώ πρέπει να δούμε όλο το φάσμα των σχετικών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην επικεντρωθούμε μόνο στην Ρωσία. Αυτές οι απαιτήσεις δεν θα αφορούν μόνο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την Ρωσία. Αυτό που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οδηγία για τα δεδομένα των επιβατών που να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες σε ενδοκοινοτικό επίπεδο. Ο κύριος Κέρκχοπ έχει δυστυχώς φύγει, αλλά θα ήθελα να απαντήσω ότι και άλλα μέλη ανέφεραν και έθιξαν το θέμα της ασφάλειας. Μπορώ να σας μιλήσω για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, ε, τα θέματα που προέκυψαν ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι καινούριο. Μετά, οι επιθέσεις στα συστήματα υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, ενέργειας. Εάν δεν υπάρχει κάποια λύση που να δίνει ασφάλεια, τότε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Κέρκοπ ανέφερε επίσης ότι και μέλη της Επιτροπής ε, πολιτικών ελευθεριών, αλλά και τα κρατημέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Και όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, πρέπει να δοθούν διασφαλίσεις, διότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Τώρα, ποιο είναι το όφελος του πακέτου αυτού για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πακέτο δεν έχει να κάνει μόνο με τα δεδομένα των επιβατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα δεδομένα των επιβατών, των επιβατών υπηκών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή τα εξέρχονται από την Ένωση. Το σύστημα δεν θα αλλάξει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει και πιο ανοιχτή και πιο ασφαλής ταυτόχρονα κίνηση των επιβατών ένα και αυξάνεται. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για τους εσωτερικούς ελέγχους και για την υποδομή. Είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για το τι ακριβώς θα χρειαστούμε και πόσα κονδύλια θα χρειαστούμε, όμως ε, πραγματικά το ερώτημά σας είναι κάτι που αφορά όλα τα κράτη-μέλη, διότι, όπως είπα, η ροή των ε, επιβατών εντός και εκτός, ε, που εισέρχονται και εξέρχονται της Ένωσης αυξάνεται κάθε χρόνο. Υπολογίζω περίπου 6 εκατομμύρια επιβάτες από τρίτες χώρες να περάσουν τα, ανατολικά σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το έξυπνο πακέτο. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα αρκετά δαπανηρό πρόγραμμα και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ που αναφέρατε, που προβλέπετε για το πρόγραμμα αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί να αγγίθει την ασφάλεια ή αν χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Αυτό δεν αφορά μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλα τα κράτη του Σέγγεν. Εάν κάθε κράτος αναλάμβανε το κόστος μόνο του, τότε το κόστος θα ήταν πολύ ψηλότερο. Η εφαρμογή των ε, συστημάτων είναι μια αναλλακτική λύση. Το πρόβλημα όμως είναι το πρόσθετο προσωπικό που θα χρειαστεί το πρόγραμμα αυτό και το κόστος του προσωπικού αυτού. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Μπερνατόνης, θα ήθελα να πω όμω ότι σχετικά με την ανατολική γειτονία αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με όλου του υπουργού και αυτό θα γίνει στι 7 και 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλου εσά, όσου ενδιαφέρεστε, να έρθετε ώστε να έχουμε μια κοινή συζήτηση. We thank also Mr. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μπερνατόνη. Παρακαλούμε τον κύριο Μπερνατόνη να συνοψίσει. Διότι έχουμε και άλλα σημεία. Δεν είναι εύκολο. να δώσει κανείς συνοπτικές απαντήσεις. Σας εκλυπαρώ το κάνετε όμως. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος μέλη της Επιτροπής για το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμά μας. Αρκετές ερωτήσεις έχουν τεθεί. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από αυτές σχετικά με αυτά που ρώτησε η κυρία Βέμπερ και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και το σχετικό πακέτο. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Θέλουμε να εξεργαστούμε και τον κανονισμό και την οδηγία. Θα είναι στην ημερήσια διάταξη του ατύπου Συμβουλίου και στην ημερήσια διάταξη της επίσημης συνεδριάσεως του Συμβουλίου των Υπουργών στο Λουξεμβούργο το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα πετύχουμε σχετικά με την οδηγία για την κατάσχεση και ανάκτηση προϊόντων εγκλήματος, εσόδων Παράνομου δραστηριότητα. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε του νομοθετήματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα στην οδηγία για την καταπολέμηση διακρίσεων. Όπως και επί ε, Ιρλανδικής Προεδρίας θα προσπαθήσουμε και εμείς να σημειωθεί η πρόοδος της ομάδας εργασίας θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις διαφωνίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη Λιθουανία και την παρέλαση Gay Pride, ποτέ δεν απαγορεύτηκε. Υπήρξε συζήτηση μεταξύ των οργανωτών και του Δήμου του Βίλνιους όσον αφορά το που θα γίνει η παρέλαση και εκδήλωση, αποφάσισε σχετικά το δικαστήριο και όπου, σαν υπουργό Δικαιοσύνης συναντώ μετακτικά με την κοινότητα των ΛΟΑΤ και τους ηγέτες της κοινότητας συζητάμε αυτά τα θέματα και η άποψή μου είναι ότι η Λιθουανία στα 20 χρόνια της ανεξαρτησίας της έχει πετύχει σημαντικές πρόοδους πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μονοπλευρή ενημέρωση για το θέμα. Ελάτε στην Λιθουανία επισκεφτείτε μας να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά τις φυλακές της CIA, συναντήθηκα με την εισηγήτρια, την κυρία Φλότρο, έγινε μια αντελεχή συζήτηση για το θέμα. Μπορώ να πω ότι η Λιθουανία έκανε τις περισσότερες έρευνες σε σχέση με τις άλλες χώρες ο Ισαγγελέφ έκανε προδικαστικές έρευνες και δεν είδαμε στοιχεία ότι υπήρξαν βασανιστήρια στο έδαφος της Λιθουανίας. Αν υπάρξουν αντικειμενικά στοιχεία για κάτι τέτοιο, ο εισαγγελέα μπορεί να ξανανοίξει την υπόθεση. Όμως αυτά τα θέματα δεν πρέπει να αξιολογούνται βάσει α, Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπίζονται νομοθετικά. Βέβαια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα, αλλά μας λείπει ο χρόνος και πιστεύω ότι απάντησα στα πιο πιεστικά ερωτήματα, στις κατεπίγουσες ερωτήσεις. Τα υπόλοιπα τα ανέφερα στην παρουσίασή μου και πιστεύω ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες και εδώ και στη Λιθουανία για να αναφερθούμε εκ νέου σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπω ότι η κυρία Μποσκούρ ήθελε μια απάντηση για την οδηγία καταπολέμησης των διακρίσεων. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στην ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Κυρία Μποσκούρ, πολύ σύντομα. Η οδηγία η κατάχρηση της αγοράς. Έθεσα ερώτημα γι' αυτό. Κατάχρηση της αγοράς. Απάντηση του Υπουργού. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στα πλαίσια της οδηγίας δεν έχουμε πρόθεση να παγώσουμε αυτό το θέμα. Θέλουμε να προωθηθεί το ζήτημα αυτό. Να προωθηθεί η οδηγία, η σχετική. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε διαπραγματεύσεις. Κυρία Μποσκούρτ, συνεχίζει ο Υπουργός να επαναλάβω για την κυρία Μποσκούρτ σαν Προεδρία Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για την οδηγία, διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς, καλώς. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συνεχίσουμε τις συζητήσεις που συνεχίζονται, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όσον αφορά την πρώτη Προεδρία Βαλτικής χώρας. Ευχαριστούμε και τους δύο υπουργούς, Μπαρασκάουσχας και Μπερνατώνης, Υπουργό Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, για αυτά που μας είπατε. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία, αποτελεσματική συνεργασία με τη Λιθουανική Προεδρία να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, να εκμεταλλευτούμε το εξάμεινο που είναι η τελική ευθεία της θητείας. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. And now, dear colleagues. Και τώρα, συνάδελφοι. Please. Rafael, hasta la próxima. Nos veremos en Vilnius, en Vilnius, Vilnius. Bye. Bye. We'll be seeing you. Bye. Zwei. Zwei. Ukrainian Thais leaving the room. Thank you all. Thank you all. Thank you all. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ ε, την προσοχή σας. Παρακαλώ προσοχή. We wave goodbye to both ministers. We thank them. Αποχαιρετούμε τους δύο υπουργού και συνεχίζουμε. Σημείο 22. Ανταλλαγή απόψεων με την και κυρία Σεσίλ Κέγκε, αξιότιμη Υπουργό Κοινωνική Ένταξη τη Ιταλία. I'm sure we all Όλοι συμφωνούμε σίγουρα πως ε, είναι τιμή μας και προνόμιό μας να έχουμε εδώ την κυρία Κίνγκε. Το άρθρο 79 της Συνδίκης Λισαβόνας αναφέρει ότι η εναρμόνιση του νόμου, η ένταξη και η ε, ε, ένταξη υπηκών τρίτων κρατών και η ευρωπαϊκή πολιτική είναι το αντικείμενό του. Η ένταξη είναι μια ε, διτή διαδικασία που καλύπτει διάφορες πτυχές, ε, απασχόληση, ε, υγεία, μεταξύ άλλων και την ε, υπηκότητα. Η Ιταλία, παρά την οικονομική κρίση, ε, εξακολουθεί να είναι χώρα αναφοράς, μία από τις ε, πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστατικό μέλος. Θέλουμε να καλωσορίσουμε την Υπουργό κυρία που θα μας ε, παρουσιάσει την πολιτική κοινωνική ένταξη της Ιταλίας. Αν επιτρέπετε κυρία Υπουργέ Κιέγγε, είμαστε πολύ, μας τιμά η παρουσία σας ανάμεσά μας. Μεγάλη χαρά, μεγάλο προνόμιο για μας να ακούσουμε άμεσα από εσά ό,τι έχετε να πείτε και πάνω απ' όλα σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συμμετάσχετε σε αυτή τη συνεδρίαση την τελευταία πριν τις στενές διακοπές τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μας τιμά η παρουσία σας, σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας και έχετε το λόγο Ευχαριστώ Ευχαριστώ τον Πρόεδρο τους βουλευτές για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε εργασίες της Επιτροπής σας που παίζει θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία που... και όσον αφορά και τα καθήκοντα που εκτελώ εγώ στην ε, Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο τον κύριο Σούλτς για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν απέναντί μου. Αυτό είναι σήμα μιας υποστήριξης και νέος νέου δρόμου, μιας νέας πολιτικής που ακολουθεί, ξεκινά να ακολουθεί η Ιταλία, αλλά είναι και σημαντικό μήνυμα για όλη την Ευρώπη. Η αναγνώριση πηγαίνει προς τον, προς την Υπουργό μου που με το διορισμό μου έκανε μια επιλογή μια προσπάθεια πολιτισμικής αλλαγής διορίζοντας επικεφαλής ενός Υπουργείου ένα άτομο που γεννήθηκε σε άλλη χώρα και που επέλεξε μια ευρωπαϊκή χώρα σαν χώρα της και σε αυτή την περίπτωση επέλεξα την Ιταλία σαν χώρα μου. Όπως γνωρίζετε, εδώ και λίγο χρόνο διορίστηκα υπουργό Ένταξης και αυτή η εντολή μου, η θητεία μου και το καθήκον αυτό το κυβερνητικό δείχνει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης στη χώρα μου και τώρα πια υπάρχει επίγνωση ότι το μεταστευτικό φαινόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαχείριση σαν κάτι κατεπήγον, αλλά χρειάζεται να κατευθυντούμε προς μια τακτική διαθρωμένη αντιμετώπιση που λαμβάνει υπόψη το άτομο σαν στοιχείο και το πλαίσιο στο οποίο διαβιώνει, που έζησε και που θα ζήσει το άτομο. Η μετανάστευση είναι ένα διαστοτικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την ιστορία αυτής της αρχής χιλιοτίας που βλέπει την Ευρώπη να μεταμορφώνεται από χώρα αποδημία σε χώρα υποδοχής είναι ένα φαινόμενο που αλλάζει τη μορφή της Υπήρου μας και το διαμορφώνει, διαμορφώνει την Ήπειρου μας σε μελλοντικές δεκαετίες. Θα πρέπει να πλησιάσουμε σε μία έννοια ένταξης υπερεθνικής. Και εννοούμε αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές που θέλουν να ισχύσουν τη διασύνδεση μεταξύ χώρας καταγωγής, χώρας προέλευσης και χώρα προορισμού μέσω διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προσπαθώντας να εντοπίσουμε θετικές λύσεις που είναι ευνοϊκές και για τις δύο πλευρές και για τους ίδιους τους μετανάστες συνεπώς. Μετανάστες που θα πρέπει να θεωρήσουμε σαν βασικό παράγοντα των πολλαπλών διαδικασιών που επηρεάζουν την οικονομία, τον πολιτισμό, την κοινωνία των χωρών υποδοχής και των χωρών καταγωγής για να επεκταθούν και σε μεγαλύτερο ακόμα επίπεδο αυτές τις επιδράσεις. Η αναγνώριση της μετανάστευσης σαν φαινόμενο διαρθρωτικό της κοινωνίας μας που μπορεί να αλλάξει τον κοινωνικό ιστό απαιτεί να ξεκινήσουν παρεμβάσεις ιδεώδεις για την συνοχή και την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, διότι με την παρουσία, διότι η παρουσία των μεταναστών εξισορροπεί τα κενά και τις ανισορροπίε συνταξιδοτικέ, δημογραφικές κλπ. Και πρέπει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει διακυβέρνηση αποτελεσματική, διακυβέρνηση του φαινομένου, τόσο ώστε να μην δημιουργηθεί κοινωνική ένταση από τη μετανάστευση, εντάσει με τον τοπικό πληθυσμό, που χρησιμοποιούνται οι εντάσει αυτέ για ιδεολογικού σκοπού. Ένα από του στόχου που θέλω να ακολουθήσω κατά τη διάρκεια τη θητεία μου είναι να αυξήσω την ευαισθητοποίηση με μεγαλύτερε μορφέ επικοινωνία, ούτω ώστε να αποφύγουμε διαστρεβλώσει, ούτω ώστε να εμποδίσουμε το ότι η μετανάστευση να μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν απειλή για την ασφάλεια. Λοιπόν, χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά την επικοινωνία, καθώς και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ορολογία σωστή μέσω συμβάσεων και συμφωνιών που ήδη υπάρχουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μοιραστούμε μια κοινή ιδέα που να είναι διαστητικά αντιληπτή, όπως είναι το αμοιβαίο συμφέρον και να υπάρχει μια ένταξη τακτική στην κοινωνία. Κάτι που τόνισε ο πρόεδρο τη Ιταλική Δημοκρατία. Και είπε, νέοι, πολι... νέοι πολίτε που έχουν επίγνωση, είναι ευαισθητοποιημένοι. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η μετανάστευση είναι, είναι ένα ενεργό στοιχείο. Όχι μόνο για την οικονομία μα, αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να είναι κινητήρα ανάπτυξη και της χώρας του. Ε, στην επικράτειά μα, οι ξένοι εργάτες γίνονται, όλο και, γίνονται και επιχειρηματίες. Σε αυτή τη νέα φάση ε, βλέπουμε αύξηση 25% σε σχέση με το 2009 των τρεχόντων λογαριασμών και των τζίρων των επιχειρήσεων που είναι η διοφυσία ε, Το δείχνουν έρευνε όσον, έγινε, όσον αφορά την οικονομική ένταξη των μεταναστών στην Ιταλία. Ελπίζουμε η οικονομική κρίση να μην επιβραδύνει αυτό το φαινόμενο που γίνεται μετανάστε επιχειρηματίε. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ χώρα προέλευση και προορισμού και θα πρέπει να υπάρχει και οργάνωση της υποδοχής και των διαδρομών ένταξης στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό θα πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα της εργασίας οι καταλυστοί, όσον αφορά υγειονομική περίθαλψη, σχολεία, κοινωνική ε, κάλυψη. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσει που δημιουργούνται. Θα πρέπει στο επίκεντρο των παρεμβάσεων να μπει το άτομο, ο άνθρωπο, ο μετανάστη, σαν δικαιούχο δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων. Αυτό είναι ο στόχο των δράσεων ε, που δρομολογώ σαν Υπουργό Ένταξη. Και από αυτού του σημείου θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Πατέρα, τον Πάπα, για την επίσκεψη που έκανε χτε στη Λαμπεντούσα και έθεσε στο επίκεντρο τη προσοχή τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, Κυρίω θέτω στο επίκεντρο των πολιτικών την αξία του ατόμου, του προσώπου. Ένα από του τομεί που θεωρώ τη θεμελιώδη σημασία είναι το σχολείο, το σχολείο αποτελεί τον ακρογωνίο λίθο της δρόμου της ένταξης. Η παρουσίαση ξένων πτυχιούχων σε διάφορους τομείς είναι ένα στοιχείο στις χώρες υποδοχής. Ενοποιητικό. Αναπτύχθηκαν διάφορα προγράμματα κατά της στην Ιταλία που έχουν σαν στόχο ε, διάφορα επίπεδα, πολιτισμούς, παραδόσεις των ομάδων προέλευσης. Θέλουμε να επεξεργαστούμε ένα σύστημα ολοκληρωμένο που να γεννάται α, να, να, να, να έχουν διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Είναι ενιαία η κουλτούρα και είναι αυτή που επικοινωνεί το κάθε άτομο και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ατόμων. Προφανώς η πρόθεση της γλώσσας που μιλάτε στον τόπο που ζει κανείς είναι η στιγμή λογής που, ε, που ε, είναι η απαρχή της ένταξης και είναι η απαρχή της επικοινωνίας αλλά και η δυνατότητα να μάθουν τα παιδιά ε, τις διάφορες γλώσσες των συμμαθητών στο σχολείο, τον πολιτισμό τους, τις παραδόσεις τους. Είμαι πεπισμένη, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία γνώσεων εμπλουτισμού πολιτισμικό. Σαν υπουργό ένταξη, λέω ότι είναι σημαντικό να συζητώ, να έχω επαφή με τον Υπουργό Παιδείας. Ήδη έχει ξεκινήσει, είναι επικοδημητικό ο διάλογο, να ξεκινήσει μια συνεργασία στου τομεί των παρεμβάσεων, ούτω ώστε το σχολείο να γίνεται ένα εργαλείο συνοχή όλο και περισσότερο και αμοιβαία γνώση και εκμάθηση. Ε, μετά εκλήθη από τον Υπουργό Εσωτερικών να συμμετάσχω στα, στις συζητήσεις τραπέζια συντονισμό για την οργάνωση της υποδοχής έναντι εκείνων ε, που ε, βγαίνουν στις παραλίες μας. Λοιπόν, είναι σημαντικό εργαλείο αυτή τη των κύριων Τραπέζη για να συντονίσουμε τι αναγκαίε παρεμβάσει βοηθεία, παροχή βοηθεία και κυρίω, και εκεί πρέπει να είναι παρόν το γραφείο μου, για να βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική αναγνώριση τη διεθνού προστασία πρέπει να ακολουθούνται σε τοπικό επίπεδο οι διάφοροι διάδρομοι ένταξη. Αυτέ οι συζητήσει απαιτούν την ενεργό συμμετοχή τη τοπική αυτοδιοίκηση, των διαφόρων διεθνών οργανισμών και των ενώσεων προστασία των μεταναστών. Ένα από του στόχου που θέλω να επιδιώξω με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Εργασία είναι να εντοπίσουμε μηχανισμού που θα πρέπει να επιτρέψουν να γνωρίζουμε από πριν τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό των προστατευμένων ούτως ώστε να ευνοούμε ε, τη συνάντηση αυτών των ανθρώπων στους εργοδότες επικαιροποιώντα και εφαρμόζοντας τις γνώσεις αυτές των δικαιούχων και να προστατεύουμε μέσω ειδικών επαγγελματικών ε, διδασκαλικών προγραμμάτων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο για την περίοδο 2014-2020 προσφέρει στα κράτη-μέλη εργαλεία όλο και πιο ευέλικτα απλά και αποτελεσματικά για τη βελτίωση των προτύπων της ένταξης και της υποδοχής. Οι πόροι είναι απαραίτητοι και θα πρέπει να συνοδεύονται όμως από πολιτικές ευρωπαϊκές διαχείρισεις με κοινέ κατευθύνσεις για να ευνοούνται διάδρομοι για την υποδοχή και την ένταξη. Η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να αντιδικοποιηθεί η καταπολέμηση εκείνων που καταχρώνται τους ε, μετανάστες. Πέρσι δέχτηκε την οδηγία για τι κυρώσει όσον αφορά του εργοδότε του 2009, ενέκρινε η Ιταλία, ώστε να τιμωρήσει εκείνου που εκμεταλλεύεται ε, του ευάλωτου μετανάστε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ε, με μηχανισμού και εργαλεία, ώστε να σταματήσουμε αυτέ τι ροέ και να καταπολεμήσουμε τι οργανώσει που κάνουν του μετανάστε νέου σκλάβους. Του εκμεταλλευτέ πρέπει να του πλήξουμε. Και θα πρέπει να έχουμε πολιτική ενιαία. Και μαζί με τι χώρε προέλευση πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική. Χρειάζεται ευρωπαϊκή η αντίληψη όσον αφορά την υποδοχή. Να τη βάλουμε στο επίκεντρο, να βάλουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού αυτή της Ευρώπης. Να βάλουμε στο επίκεντρο το άτομο του όλου προβληματισμού. Λοιπόν, καλούμε να συνεχίσω στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας και διάκρισης. Η Ιταλία έχει ειδικέ νομοθεσίες, ειδικού νόμους όσον αφορά τα θέματα αυτά και οι συνεργάτες μου εξεργάζονται νέα εργαλεία και νομοθετικού περιεχομένου για να εμποδιστεί ή ε, πρόκληση για πράξεις ρατσιστικές και ίσως και μέσω των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας. Ο ρατσισμός πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταπολεμηθεί πολιτισμικά. Αυτό αντιπροσωπεύει την βασική αρχή των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και πρέπει να προωθηθούν. Λοιπόν, η διαδρομή, η πολιτισμική, είναι αυτή που ακολουθώ και όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής της εθνικής, όσον αφορά την ένταξη των Ρωμά. Θέλουμε να έχουμε προγραμματισμό βάσει τη αποφάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτού του πληθυσμού. Αν η μετανάστευση δίνει δυνατότητε και πόρου, θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα. Να δίνουν ευκαιρίε για του μετανάστε, για την κοινωνικό όστο και θα πρέπει να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία τη ένταξη. Ε, είναι νέα, θα, νέα υπηκότητα μέσω τη μετανάστευση. Από την αρχή το έθεσα σαν στόχο, από όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Νέα ηθαγένεια όπου όλοι μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Μπορούν μέσω νομίμων διαδρομών να υλοποιούν τις, ε, τα οράματά τους. Θα πρέπει ο πολίτης να είναι στο επίκεντρο και θα πρέπει να προβλέπεται και συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των μεταναστών. Σήμερα γίνεται πολιτική συζήτηση στη χώρα. Έχει οριμάσει η συζήτηση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις φυσικές συνέπειες των πολιτικών ένταξης χρειάζεται κοινό προβληματισμό που να μπορεί να οδηγήσει σε νέα νομοθεσία όσον αφορά την ηθαγένεια, την υπηκότητα. Στο Κοινοβούλιο τη Ιταλία έχουν κατατεθεί πάνω από 20 προτάσει νομοσχεδίων και τα περισσότερε βασίζονται σε κοινού στοιχείου. Να αναγνωριθεί κατά κάποιο τρόπο το καθεστώ σε εκείνο που γεννάται στην Ιταλία και αποκτά ε, την γλώσσα και τον πολιτισμό. Προστίθεται μετά ε, ε, και οι Ιταλοί στο εξωτερικό. Η δυνατότητα να μπορούν να εργαστούν και όσον αφορά το θέμα τη υπηκότητα με του Ιταλού που είναι στο εξωτερικό. Ξεκίνησε πρώτη σημαντικό αποτέλεσμα όσον αφορά την απλούστευση, προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών χορήγηση τη υπηκότητα, χάρη στην πρωτοβουλία του δικού μου Υπουργείου. Στο, στη διακή, στο νομοσχέδιο για την απλούστευση υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη, άμεση διάταξη, για να αποφύγεται ότι αυτό που γεννήθηκε από γονεί που νόμιμα διαμένουν και είναι πάνω από 18 να, να μην να στερείται την υπηκότητα λόγω εμποδίων γραφειοκρατικών που, για τα οποία δεν φταίει ε. αυτό. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα. Το χύτερο δυνατόν πρέπει να καλυφθούν τα κενά, κατά την άποψή μου, ε, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα συνοδευτικά μέτρα που είναι τα αποτελεσματικότερα για να ενισχυθεί η ε, συνεργασία και ανάπτυξη. Να γίνει ενεργό ο μετανάστης στη χώρα μας. Και για τη χώρα προέλευσης και για τη χώρα υποδοχής. Μόνο μέσω μία κοινή διαδρομής, συνεχούς διαλόγου και ανανομένης επίγνωσης και γνωστοποίηση μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν εχθροί και δεν υπάρχουν άλλοι. Πρέπει να έχουμε πολιτικές υποδοχής, ένταξης και συμπερίληψης, ούτω ώστε σε οικονομικά δύσκολε περιόδους όπω είναι η παρούσα να δημιουργήσουμε νέε ευκαιρίε για ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Grazie lei. Άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ που ανταποκριθείτε καταθετικά στην πρόσκλησή μας και σας ευχαριστώ που επικεντρώσατε την παρέμβασή σας επί των σημαντικών σημείων για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ελευθερία, δικαιοσύνη, ε, θέματα εσωτερικών. Έχουμε έναν κατάλογο που δεν είναι ε, σύντομος, μελών που θέλουν να μιλήσουν. Προτείνω λοιπόν ε, να είστε λακωνικοί, να έχετε υπόψη πριν πάρετε το λόγο αυτό να προλάβουμε, διότι δεν είναι το τελευταίο σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, τη σημερινή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η κυρία Ματιέ, έχετε το λόγο. Ε, με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε, Υπουργέ, εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα είμαι σύντομη. Άκουσα με προσοχή την ομιλία σας ένταξη, επικοινωνία, συνοχή, διαχείριση της υποδοχής ήταν λέξεις οι οποίες ε, επανερχόντουσαν. Πρόκειται για μια ομιλία με, πολύ, με πολλές ανθρώπινες ε, και ανθρωπιστικές αναφορές. Μίλησατε επίσης και για δικαιώματα και υποχρεώσεις προκειμένου να γίνει επιτυχής η ένταξη. Ευθύνες έχουν όλες οι πλευρές. Εσείς ε, στο μυαλό σας έχετε τη διαχείριση της μετανάστευσης με ένα τρόπο πραγματικά ε, που θα αποφύγει το να φτάσουμε στα άκρα που έχουμε φτάσει. Μιλήσατε για την εκπαίδευση των μεταναστών, μιλήσατε για την επιτυχία της ένταξης μέσω συγκεκριμένων βημάτων. Ε, μιλήσατε για τη σχέση με τις επιχειρήσεις, με τη σχέση με τον τραπεζικό κόσμο, ε, με συγκεκριμένα μέτρα ε, επιχειρηματικά και στον τραπεζικό τομέα που θα βοηθήσουν την ένταξή τους. Έτσι ώστε οι μετανάστες να αισθάνονται αποδεκτοί πρέπει να εργάζονται Μιλήσατε για επικοινωνία, μιλήσατε για ε, γνώση της γλώσσας. Στην ομαρχία των Βοσγίων ξεκινήσαμε μια ε, διαδικασία ε, νομοποίησης μέσω ε, μιας υποδοχής από τις κατάλληλες υπηρεσίες της νομαρχίας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εκμάθηση της γλώσσας μας είναι πολύ σημαντική και για τους μετανάστες αλλά και για τον τόπιο πληθυσμό έτσι ώστε πραγματικά αυτοί οι μετανάστες να ενταχθούν και να αποφευθούν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Μας αναφέρατε ότι ετοιμάζετε διάφορα νομοσχέδια αλλά ειλικρινά μπορούμε να έχουμε βουνά νομοθεσίας στην πραγματικότητα όμως οι νόμοι δεν λύνουν τα προβλήματα όπως αυτά της ξενοφοβίας, το ξέρετε πολύ καλά. Η καλή ένταξη, η καλή επικοινωνία ανάμεσα στο μετανάστη και τον τόπιο πληθυσμό είναι αυτά που λύνουν το πρόβλημα. Καλό κουράγιο και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ελπίζω ότι θα, καταφέρετε, θα τα καταφέρετε στην Ιταλία. Ωραία. Ο λόγος στην κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την Υπουργό για το σαφές όραμα που έχει, για την τόλμη της και τη γενναιότητά της. που φαίνεται στις προτάσεις που υποβάλλει. Πολύ συχνά οι πολιτικοί περιορίζονται στο λαϊκισμό. Σε ό,τι φορά την ένταξη, έχω την εντύπωση ξεκινούμε συνεχώς από το μηδέν, σαν να κάνουμε γύρους γύρω από τον εαυτό μας. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες Κοινωνική ένταξη. Να σα πω το εξή. εγώ είμαι κόρη μεταναστών. Στις κάτω χώρε. Και εδώ εκπροσωπώ τις κάτω χώρε. Αλλά συχνά θεωρούμε ακόμα μετανάστρια. Πότε τελικά κάποιος πάβει να είναι μετανάστης και έχει ενταχθεί πλήρως. Γιατί διαιωνίζεται ο χαρακτηρισμός του μετανάστη πολύ συχνά. Θα έπρεπε να τελειώνει αυτό στην Ευρώπη. Πώς μέσω της έννοιας της ε, ε Υπάρχουν πολλές ιδέες όπως της ε, μπλε κάρτας κλπ. Αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το διχασμό ανάμεσα σε μετανάστες και Ευρωπαίους. Ο κ. Γιακολίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό που δέχτηκε χωρίς δισταγμούς ε, την πρόσκληση της Επιτροπής μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, τις περασμένες ημέρες, κυρία Υπουργέ, εγκρίναμε ένα πακέτο που επανακαθορίζει το καθεστώς του ασύλου στην Ευρώπη. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ένας είναι ο, ο, κανονισμός του Δουβλίνου, ένας από, τα, από τις πτυχές, που είναι επικεφαλής όλων των θεμάτων που αφορούν τη διαμονή του πρόσφυγα κάποιου που δεν μπορεί να μείνει πλέον στην χώρα προέλευση και μετά πρέπει να υποστηριχθεί αυτό ο άνθρωπος και να προστατευτεί. Πρόσφατα οι Υπουργοί Εσωτερικών είπαν ότι ένα από του πρώτου στόχου, ο Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών, είπε ότι, ε, θα είναι επανεξετάσει τον κανονισμό του Δουβλίνου. Προσπαθεί να κάνει να καταλάβουμε τα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται ευθύνη να μοιραστεί μεταξύ κρατών μελών, ευθύνη έναντι των μεταναστευτικών ροών είτε είναι νόμιμες ηρωές ή περισσότερο όταν είναι παράνομες ηρωές. Θα, θα επανεξεταστεί αυτό, θα κάνει κάτι γι' αυτό ο υπουργό. Χθε ο Πάπας ε, Φραγκίσκος, όπως υπενθυμίσατε σωστά, μετέβη εις Λαμπεντούσαν και φώτισε αυτό το μονοπάτι της ελευθερίας που αφορά τους πρόσφυγες, τους μετανάστες που καταφθάνουν εκεί. Ήταν μια ημέρα πολύ έντονη, μεγάλη έντασης έναντι των μεταναστών ανεξάρτητα της θρησκείας τους ε, και αυτό είναι κάτι μας γεμίζει χαρά. Αναφερθήκατε σε κοινού κανόνες για όλους τους μετανάστες αναφερόμενοι και στην ε, απόκτηση τσιπικότητας. Πώς, γιου σόλε, ε, ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αναγνωρίζετε αυτό το καθεστώς. Εμείς υπέρ ενός πολιτισμού κουλτούρας ένταξης και υποδοχής για να αντιταχθούμε σε κάθε διάκριση. Και χαιρόμαστε που μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ιταλική κυβέρνηση και με τι άλλε κυβερνήσει, ούτως ώστε να θεσπίσουμε κοινού κανόνε που στηρίζουμε όλοι, όλα τα κράτη-μέλη. Ξεκινώντα από την υπόθεση ότι υπάρχει πραγματική αυθεντική αλληλεγγύη έναντι κυρίω των χωρών του Νότου, όπω η δική μα χώρα που υποφέρουν από πολύ μεγάλες, τρομερές μεταναστευτικές πιέσεις. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνη. Ε, κυρία Ρομέρο Λόπες. Και εγώ θα ήθελα να δω συνέχεια σε αυτά που είπε ο κύριος Γιακολίνο λέγοντας ότι ε, χαίρομαι που η Ιταλική κυβέρνηση σκέφτεται τι, κάνει, τι θα κάνει ήδη με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Μόλις τον εγκρίναμε εδώ ε, και έχουν αργήσει οι κυβερνήσει του Νότου να αντιληφθούν το τι συμβαίνει με τον οργανισμό του Βλήνου. Μακάρι οι, όλες οι κυβερνήσεις του Νότου να είχαν καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί ο αριθμός των ετούντων άσυλο μέσω αυτών των χωρών θα είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει να παραμείνουν εκεί. Ε, και καταλαβαίνετε ότι με την οικονομική κρίση αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Ε, χαιρόμαστε για την επίσκεψη του Πάπα Φρανσίσκου αλλά είναι ευθύνη των κρατών μελών να διοργανώσουν σωστά και με καλές συνθήκες τα, ε, τους χώρους κράτησης ε, όπως αυτός της Λαμπεντούσα. Απ' την άλλη μεριά είναι σημαντική η διμερής συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, για παράδειγμα την Ισία ή Λιβύη σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Γιατί πολλά ατυχήματα στη θάλασσα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν είχατε συνεργαστεί ε, με τη Λιβύη και την Τινησία όπως η Ισπανία έχει συνεργαστεί με το Μαρόκο. Και επιτέλους αρχίζουμε και μιλάμε για τη μετανάστευση με διαφορετικούς τρόπους, όχι για παράνομη μετανάστευση, ε, μάλλον όχι μετανάστευση συνδεδεμένη με, την, ε, με το έγκλημα, αλλά με ένα τρόπο διαφορετικό όπως αυτός που ε, έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Η μετανάστευση αποτελεί πλούτο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας, γιατί εδώ και πολύ καιρό ακούμε τη μετανάστευση συνδεδεμένη μόνο με το έγκλημα και την παρανομία. Όμως ε, οι μετανάστες οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι πλούτος ε, και έχουμε πολλά πολιτικά μέσα στη διάθεσή μας για την ένταξη των μεταναστών. Εσείς αναφέρατε ορισμένα από αυτά. Ίσως θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε σε ορισμένα. Συνεργασία με τους ε, δήμους και τις κοινότητες των χωρών προέλευσης. Ε, οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές, ένας θεσμός καινούριος και ε, πολύ ωφέλιμος. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε την παρανομία και τα υπόλοιπα προβλήματα. Η κυρία είναι Αντζελίλη. Επαναλαμβάνω, θυμηθείτε το χρόνο. E Ευχαριστώ. και την κυρία Υπουργό που ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάποια σκέψη και ερώτηση. Πιστεύω ότι καλά κάνατε που είπατε ότι τα θέματα που άπτονται της μεταναστεύσεως δεν μπορούν να μπουν να εξετάζονται κατεπήγοντα. Όπως είπατε χρειάζεται ένα πρόγραμμα, σαφείς κανόνες, δικαιώματα, υποχρεώσεις Σωστά το είπατε και επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα πιο ευάλωτα άτομα και ιδιαίτερα τα παιδιά. Και πολλοί αναφερθήκατε στις έννοιες της ένταξης και της αλληλεγγύης. Προφανώς μοιράζομαι και εγώ την ίδια προσέγγιση. Όμως πρέπει να σκεφτούμε την έννοια της ένταξης, της αλληλεγγύης και του, της κοινή προσέγγισης, του μοιράσματο. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ίσως θα περίμενα, πώς να το πω, από την πλευρά σας, μία έκκληση να ακούσω. Είστε Ιταλίδα υπουργό, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία έκκληση για την αλληλεγγύη όπως αποκαλείται, την ενδοκινοτική. Είναι μία έννοια που δυστυχώς μπάζει νερά από παντού. Και αυτές τις μέρες Στη Λαμπεντούσα, παραδείγματο χάρη, δεν πήγε μόνο ο Πάπας Φραγκίσκο, αλλά έγιναν και από. Ε, βγήκανε και άτομα, κατέφθασαν άτομα, πρόσφυγες, στις γνωστές συνθήκες κατέφθασαν, απελπισμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς, ε, μεταξύ Μάλτας και Λαμπετούσας ε, ρίχνεται το μπαλάκι της ευθύνης. Καμιά φορά παίζει με την Ιταλία, την Ισπανία, με την Ελλάδα, την Ισπανία κλπ. Το πρόβλημα είναι μόνο των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης. Όταν μιλάμε λοιπόν για μοίρασμα των ευθυνών και αλληλεγγύη και επέκρινα πολύ το θέμα εγώ όσον αφορά την έγκριση του πακέτου μετανάστευσης. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κοινή προσέγγιση, για αλληλεγγύη, για μοίρασμα της αλληλεγγύης, ουσιαστικά μιλάμε για μια αλληλεγγύη που είναι στις πλάτες των χωρών που πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατεπίγουσα ανάγκη, την κατεπίγουσα κατάσταση. Λοιπόν, κάποιες χώρε έχουν δικαιώματα και καθήκοντα και άλλες χώρες έχουν μόνο δικαιώματα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό θα ήθελα να στείλετε μία έκκληση. Διαφορετικά η λιλεγγύη γίνεται κενό γράμμα και απλώς ε, ρητορικό σχήμα. Ευχαριστώ η κυρία Κώστα. Η ε, κυρία Υπουργέ, μεγάλη τιμή και ε, μας δημιουργεί συναισθήματα συγκίνηση που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εξέφρασε αλληλεγγύη το θέμα και σαν Ιταλίδα Ευρωβουλευτή, χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι η παρουσία σας έχει συμβολική σημασία και πολιτική σημασία που δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε από την Ιταλία ούτε από την Ευρώπη αυτό το νόημα. Όσον αφορά αυτά που είπατε, τα συμφωνώ και σα υποστηρίζω και τα εκτιμώ αυτά που είπατε. Ε, πιστεύω ότι το αίτημα που θέσατε και αναφέρατε στην παρέμβασή σας ε, αφορούσε μάλλον, μιλήσατε και αυτά που κάνει η χώρα μας και όσον αφορά αυτό το ζήτημα ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρει μια χαμένη αλληλεγγύη, δικαιοσύνη ε, και σεβασμό του ατόμου, όπως είπατε, στο πρόσωπο του μετανάστου. Χρειάζεται πιο προσεκτική τοποθέτηση διάδρασης περισσότερο από ότι ένταξης. Και υπάρχει διαπολιτισμικός παράγον που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες της πολιτισμικές της ένταξης. Πιστεύω λοιπόν ότι και η χθεσινή επίσκεψη του Πάπα που δεν μίλησε μόνο στους χριστιανούς αλλά μίλησε στους πιστούς και στους μη πιστούς και στους Ευρωπαίους και είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε μια, ένα χαμένο αίσθημα αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και να κινηθούμε κατά τη διαφορία στον αφορά αυτές τις αποβάσεις. 20.000 άνθρωποι πνίγηκαν πιθανότατα στη Μεσόγειο. Τρία σημαντικά σημεία να ε, θέλω να υπογραμμίσω και θέλω θέση σας. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι σε αντίφαση με αυτή την πολιτική της αλληλεγγύης και της υποδοχής της νόμης συμπεριφοράς και της αλληλεγγύης, το γεγονός ότι υπάρχει το αδίκημα ε, της παρανομίας ε, όσον αφορά ε, την παραμονή στη χώρα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Κάποιοι που γίνονται παράνομοι για θέματα γραφειοκρατικά γίνονται παράνομοι και μπαίνουν στο χώρο του αδικήματος και αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Το θέμα της υπηκότητας που θε, σαν ιταλικό ζήτημα στα πλαίσια νομοθεσία έχει και αντίκτυπο ευρωπαϊκό. Διότι ένα παιδί που γεννάται σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, έναν τη Ιταλία τουλάχιστον θεωρείται ε, Ευρωπαίος πολίτης, έχει δικαιώματα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, είναι η, αν η ευρωπαϊκή υπηκότητα συμπληρώνει την εθνική εισαγένεια, ε, σημαίνει ότι υπάρχει και πρόβλημα έναν της Ευρώπης η χορήγηση υπηκότητας. Το είπε συνάδελφος Ρομέρο και η κυρία Αντζελίλη το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτικών που επιθυμείτε, αυτό είναι ενδιαφέρον σημείο. Θέλουμε να έχουμε ε, από την πλευρά σα ε, περισσότερε προτάσει προ αυτή την κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη, πιστεύω ότι είναι σωστό που έγινε αυτό που κάναμε, διμερείς συμφωνίε με την Ισία. Όμω άλλαξε κάπω το πλαίσιο, το ξέρουμε, στη Βόρεια Αφρική. Όμω πιστεύω ότι η δική μα πρόταση των βουλευτών και τη ομάδα μου ήταν πάντα αυτή. Να έχουμε διμερεί συμφωνίε Ευρώπη με αυτέ τι χώρε και να μην αφήσουμε μόνο τι χώρε της ε, ε, Μεσογείου ε, να κινούνται σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ κυρία Κώστα, η κυρία Κέλλερ. Thank you very... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ που ήρθατε. Δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία συχνά, αυτή την ευχαρίστηση να έχουμε έναν υπουργό που δεν είναι κάποιας χώρας που έχει την προεθρία. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σε αυτή την επιτροπή έχουμε την τύχη να βλέπουμε άτομα που δεν βλέπουμε συχνά και αυτό δείχνει και πόσο ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσία σας, η προσέλευση. Πιστεύω πως είναι πιο πραγματιστική η προσέγγιση αυτή που μας παρουσιάσατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και σας εύχομαι καλή τύχη με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στην Ιταλία. Επίσης συμφωνώ με όλα όσα είπατε για το ρατσισμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό παντού, στην κοινωνία, στην πολιτική, στον πολιτισμό. Θα χρειαστούν πολλά βήματα και όχι μόνο νόμοι για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό. Και πιστεύω πως είναι σημαντικό να μην συγχαίουμε την ένταξη και την με την καταπολέμηση του ρατσισμού, διότι το, η καταπολέμηση του ρατσισμού δεν είναι έργο των μεταναστών, δεν είναι κάτι, είναι κάτι που θα επιληθεί, δεν είναι μάλλον κάτι που θα επιληθεί όταν έχουν ενταχθεί όλοι. Όχι, αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δυστυχώ, ο ρατσισμό δεν κοιτάζει το παρελθόν του κάθε ατόμου. Ο ρατσισμό πρέπει να καταπολεμηθεί παγκόσμια, σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εκφάνσεις του. Τώρα μια ερώτηση ως υπουργό Ένταξης. Ε, να σας ρωτήσω πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στην υλοποίηση του προγράμματός σας ε, μέσω προγραμμάτων, μέσω απόκτησης δεξιοτήτων. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θέλατε εσείς να δείτε Μέχρι τώρα το μόνο που κάνουμε είναι να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Ποια είναι λοιπόν τα βήματα που πιστεύετε πως θα έπρεπε να λάβουμε για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ρωμέγο Δεφοντάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε Υπουργέ. Σε πολλά σημεία συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή πρέπει να κλείξουμε την εκμετάλλευση των μεταναστών. Διότι πολλές φορές πρόκειται περί εκμεταλλεύσεως αυτό που διαπιστώνουμε και είναι τεράστιο κακό για την ανθρωπότητα. Προφανώς, ίσως οι πολιτικές με τις οποίες θέλετε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα ή θέλουμε είναι διαφορετικές. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, σωστά είπατε ότι οι μετανάστες για να ενταχθούν πρέπει να έχουν δουλειά, στέγαση, περίθαλψη, υγειονομική. Ξέρετε ότι περνάμε πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές και ξέρετε ότι στην Ευρώπη έχουμε περίπου 26 εκατομμύρια ανέργους. Στην Ιταλία αυξάνεται η ανεργία. Μιλήσατε για ξένους επιχειρηματίες. Εγώ προέρχομαι το Βένετο. Οι επιχειρηματίες στο Βένετο αντί να εργάζονται πρέπει να αυτοκτονούν λόγω του Ιταλικού κράτους και των φόρων που βάλει το Ιταλικό κράτος. Και πολλοί νέοι από το Βένετο μεταναστεύουν. Μέχρι τη δεκαετία του 60 είχαμε μετανάστευση και ξαναρχίσει αυτή τη δικασία Από τη δεκαετία του 60 έχει ξαναρχίσει. Πώ μπορεί να ενταχθεί η μετανάστευση και ο μετανάστη όταν υπάρχουν δυστυχώ αυτά τα οικονομικά προβλήματα και η ανεργία για εκείνου που ζουν επιτόπου τόπου. Εάν δεν υπάρχει δουλειά είναι δύσκολη η ένταξη. Εγώ αυτό πιστεύω. Ίσως, τι να πω, αυτή είναι η άποψή μου. Άκουσα που λέγατε ότι στην κοινωνία υπάρχουν ανισορροπίε, Ανισορροπίε που οφείλονται σε ένα πληθυσμό που ε, γυράσκει. Πέρα από το γεγονό ότι χρειάζεται αντιστάθμιση των αυτών ανισορροπιών των δημογραφικών μέσω μετανάστευση, μήπω κάτι πρέπει να γίνει για τι πολιτικέ τη οικογένεια, ούτω ώστε οι οικογένειε στην Ιταλία να έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν καλύτερα τα παιδιά του, Ξέρω εγώ να μειωθούν κάποιοι φόροι, να βοηθούν οι πολίτεχνες οικογένειες, να βοηθηθούν. Τέλος, σωστά, αναφερθήκατε σε θέματα κουλτούρας, νοτροπίας. Είπατε ότι υπάρχουν περισσότεροι πολιτισμοί που πρέπει να ταιριάξουν μεταξύ τους. Και σωστό. Και είναι η τελευταία ερώτηση. Πώς τίθεστε έναντι των νοοτροπιών που καταφθάνουν σε εμά χάρη στη μετανάστευση. Το χειρότερο κομμάτι της μετανάστευσης. Νοοτροπίες που φέρνουν την εφαρμογή της αρία. Ε, θεωρείτε ότι αυτές οι μορφές, αυτές οι νοοτροπίες ε, έχουν νομιμότητα, μπορούν να εφαρμοστούν στις ε, περιοχές μας. Ευχαριστώ, κύριος Ροντζούλη. Κυρία Ροντζούλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Και εγώ εν μέρη συμφωνώ με αυτά που είπατε και ήθελα να εκφράσω κάποιες σχέσεις. Στην ακρόασή σας, αυτά που είπατε, αναφέρατε αυτά από το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε Δεν πέρασε να με αυτό το μήνυμα μεγάλου ανθρωπισμού και αλληλεγγύης του Πάπα με τις πολιτικές απαιτήσει που έχει μια χώρα όπως η Ιταλία. Ειλικρινά σας λέω και ζητώ συγγνώμη. Ίσως, ίσως είμαι η μόνη σκληρή παρέμβαση μέχρι τώρα. Σαν καθολική και σαν γυναίκα των θεσμικών οργάνων απογοητεύομαι όταν βλέπω πως κάποια λόγια του Πάπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδεολογικούς σκοπούς. Όλοι μας, πιστεύω καν, μηδενός αποκλειωμένου, εξαιρουμένου, προσεύχηθηκε και προσεύχεται για εκείνους που χάνουν τη ζωή στη θάλασσα. Όμως, οι απαιτήσει υπάρχουν απαιτήσει για την ασφάλεια μιας χώρας και δεν θα πρέπει να έχουν πιο μειονεκτική θέση. Εκτενώς αναφερθήκατε στη λέξη μετανάστης. Πολύ συχνά αναφέρατε αυτή την έννοια. Και ποτέ τη λέξη νομιμότητα σχεδόν. Βελτίωση της πολιτικής υποδοχής όσο με αφορά δεν σημαίνει μη ρύθμιση, μη νομιμοποίηση, μη νομοθέτηση. Και κυρίως δεν πρέπει να ε, παγρυπνούμε λιγότερο. Ε, κλείνω με κάτι που υπόθηκε από τους συναδέλφους, αλλά το επαναλαμβάνω και εγώ. Εδώ και δύο χρόνια, σε αυτό το κοινοβούλιο, η Ιταλία βρέθηκε απομονωμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό των μεταναστών στη Λαμπεντούσα. Η Λαμπεντούσα θεωρήθηκε σαν ένα κομμάτι, σαν σκολικοειδής απόφυση της Ιταλίας και όχι σαν νότια ακτή της Ευρώπης. Και κλείνω με μια ερώτηση. Έφτασα στα όρια μου, ίσως το κατάλαβα. Το κατάλαβα και από τη σημερινή συνέντευξή σα. Είπατε ότι να θέσουμε την ασφάλεια σε πρώτη θέση στην αντιμετώπιση των θεμάτων τη μετανάστευση προϋποθέτει έναν τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου της μετανάστευσης που είναι απόμακρο από τον τρόπο με τον οποίο τον λαμβάνομαι εγώ. Και μετά συνεχίσατε λέγοντα ότι προτείνεται την, ε, την ένταξη, την υποδοχή σαν προσέγγιση. Ακούσαμε ένταξη, υποδοχή κλπ. Αλλά δεν κατάλαβα σαν πώς η κυρία Υπουργό προτίθεται να συμφιλιώσει όλα αυτά με την νομιμότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορκέτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, μας παρουσιάσατε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό και σκοπό την υλοποίηση αυτό που δεν κατάφερε να υλοποιήσει η χώρα μας και ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Σοβαρό πρόγραμμα ένταξης. Εγώ σας ε, ε, απευθύνω θερμότατες ευχές, διότι θα ήταν πολύ σημαντικό να πετύχετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Από αυτή την ε, άποψη, κανείς όπως εμάς και το δικό μας πολιτικό κόμμα δεν θα αφισβητούσε ότι πρέπει να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Η αμφιβολία είναι σαν αυτό το δρόμο που θα ακολουθηθεί για το σκοπό. και τα σημεία αναφοράς. Παραθέτω αφορά σημεία σαφώς, που αναγνωρίζω και ότι εσείς ήσασταν ειλικρινείς και ήσασταν και ευγενέστατοι έναντι εκείνων που σας επετέθησαν. Αλλά έχω να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλετε να μιλάτε για τους παρανόμους, τους κρυφούς. Αλλά γνωρίζετε, διότι είσαστε ευφυής άνθρωπος, ότι πολλά άτομα ή κάποια άτομα έρχονται στη χώρα μας και στις ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα μας τουλάχιστον όσον αφορά, όχι για να βρουν δουλειά ή για να λύσουν ένα πρόβλημα και πείνα ίσως, αλλά με πρόθεση να διαπράξουν εγκλήματα, δικήματα, όχι μόνο από την Αφρική, αλλά και από άλλα μέρη της Ευρώπης. Ε, λοιπόν, και αυτούς πώς συμπεριφερόμαστε, τους, τους διώχνουμε, τους απελάβνουμε, όπως κάνει η χώρα ε, ε, προέλευσης που είναι πολύ σοβαρή έναντι των παρανόμων. Και ο Πάπας μίλησε για σκοτεινούς σχεδιασμού που ευνοούν αυτά τα διεθνή δράματα. Εγώ σας ρωτώ, συμφωνείτε όταν λέμε ότι ένα δίκημα κατά ανθρωπότητα είναι να, έχουν, να κάνει τους ανθρώπους ριζοσπαστικού, να ακολουθούν ακραίε θέσει. Σας φαντάζομαι εγώ μια κοπερίτσα 15, χρόνια, 15 χρονών που τη φέρανε την φέρανε στην πόλη και κυκλοφορούσε στους δρόμους και έτσι χωρίς να την προσέχει κανένας. Εγώ ήμουν ρατσιστής που είπα στις αρχές να φροντίσουν αυτό το κοριτσάκι που ήταν 15 χρονών. Ξέρετε ότι πολλές οργανώσεις όπως τη χώρα μου λένε ότι παρέχουν βοήθεια αλλά τελικά κερδοσκοπούν όσον αφορά τη βοήθεια που δίνουν στους μετανάστες. Έχετε σαν υπουργό ε, όλα τα μέσα ούτως ώστε να ρίξετε φως σε αυτό. Ε, Μετσόλα. Η κυρία Μετσόλα, ευχαριστώ ε, Υπουργέ, εκτιμώ την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Ο, Ο Πάπας χθες είπε ξεχάσαμε να, κρέμε, να κλέμε. Ε, αυτό είναι ισχύει για όλους μας στη Μεσόγειο ε, και μας ε, ξύπνησε. Ελπίζω να ξύπνησε και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καημός των ανθρώπων που διασχίζουν τη Μεσόγειο δεν πρέπει να αγνοηθεί και θα πρέπει να χάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Μαζί όμως με αυτό το θέμα, παράλληλα, υπάρχει και το θέμα της ελεγγύης. με ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται πάνω-πάνω στην μέση διάταξη στη χώρα μου, τη Μάλτα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς οι πολιτικοί αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, όλη τη μέρα. Εμείς ε, στη Μάλτα θεωρούμε ότι έχουμε αφαιθεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα μόνοι μας. Στο πακέτο που υιοθετήθηκε τον περασμένο μήνα ε, ε, διατηρεί τα προβλήματα που είχαμε με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Και πιστεύουμε ότι παρόλο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την αλληλεγγύη του επανειλημμένως σε χώρες όπως η δική μου, για παράδειγμα σε θέματα μετεγκατάστασης, αυτή η αλληλεγγύη δεν επιδείχθηκε από πλευρά του Συμβουλίου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο εμείς να πάμε σπίτι και να πούμε στους ανθρώπους εκεί ότι από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μας ακούει κανείς. Και είναι δύσκολο να τους εξηγήσουμε το ότι κυρίως κυβερνήσεις άλλων κρατών ε, αποφεύγουν να μας βοηθήσουν με ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, που είστε παρούσα. Ευχαριστώ για αυτό που κάνετε και όπως το κάνετε στη χώρα μας θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις. Όχι ερώτηση. Αναφερθήκατε εκτενώς στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Θα ήθελα να αντιστρέψω την έννοια το πρόβλημα είναι των μεταναστών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε πολύ στην επίσκεψη του Πάπα. Αναφερθήκατε και με ένα κριτικό πνεύμα. Είναι θρησκευτικό ηγέτη. Πάει σε μια κοινότητα ο Πάπα, εκφράζει τη δική του αντίληψη βάσει τη ιδιότητά του και αυτό που εκπροσωπεί. Μίλησε πολύ για αλληλεγγύη ο Πάπα. Η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο μία έννοια του Πάπα. Αλληλεγγύη είναι μία έννοια θεμελιώδη τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εδράζεται επί τη αλληλεγγύη. Λοιπόν, τι σημαίνει να είναι κανεί αλληλέγγυο. Σημαίνει ότι αν βρούμε ένα άτομο στη θάλασσα που πνίγεται, να το ρωτήσουμε αν έχει πρώτα διαβατήριο και αν φτάνει νόμιμα ή αν φτάνει παράνομα. Ή Εκείνοι που φτάνουν στην επικράτειά μας πρέπει απαραίτητα να θεωρηθούν σαν παράνομοι και να αντιμετωπίζονται τέτοιο τρόπος στα κέντρα κράτησης, διοικητικής κράτησης που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης διότι δεν έχουν καμία βάση νομική. Ή η Λαμπεντούσα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί αντιδρά διαφορετικά σήμερα σε σχέση με το πώς αντιδρούσε πριν από καιρό. Όταν είχε πλημμυρίσει από άτομα η ε, Λαμπεντούσα και οι ντόπιοι έπρεπε να αντιδράσουν γιατί δεν μπορούσαν καν να σταθούν. Πώς σήμερα που φτάνουν συνέχεια πρόσφυγες ο ένας μετά τον άλλο οι βάρκες το νησί της Λαμπεντούσα δεν αντιμετωπίζει τις συνθήκες. Ίσως γιατί το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο δεν έχουν εγκαταληφθεί ε, να μην μαζεύονται σε τόπους ε, και να στριμώχονται οι άνθρωποι αυτοί και να αντιδράσουν. Πέρσι πήγαμε με την επιτροπή μας στη Λαμπεντούσα, επισκεφτήκαμε άλλα κέντρα υποδοχής, ε, άλλα κέντρα κράτησης, όπως τα έχω ορίσει, και είδαμε πως όταν φτάνουν στην Ιταλία αυτά τα άτομα γίνονται μόνο αριθμοί. Καμιά φορά δεν είναι καν νούμερα αυτοί οι άνθρωποι, διότι απλούστατα πρέπει να φύγουν και δεν έχουν κάνει τη δυνατότητα να το κάνουν, να φύγουν. Εμείς πρώτοι επικαλούμεθα τους κανόνες. Οι ίδιοι μετανάστες επικαλούνται τους κανόνες για να μπορούν να ζήσουν σε διαφορετική κατάσταση. Αυτή η αλληλεγγύη που η Ευρώπη, όχι μόνο η Ιταλία, που η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να έχει έναντι αυτών. Ευχαριστώ κύριο Κλέης. Eh, eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Η πραγματικότητα εδώ, σε αυτή τη χώρα, δείχνει ότι η δυσκολία ένταξης προκύπτει πολύ συχνά από την έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας των μεταναστών στη χώρα τους. Για παράδειγμα, όταν προέρχονται από μια χώρα που εφαρμόζει τη Σαρία και επιθυμούν να την εφαρμόσουν και εδώ στην Ευρώπη, όταν προέρχονται από ένα περιβάλλον πολυγαμίας ε, ή ακροτηριασμού γεννητικών οργάνων, πώς είναι δυνατόν να κλείσουμε τα μάτια σε όλα αυτά. Πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και των παιδιών τους. Αναφερθήκατε σε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Θεωρείται υποχρέωση των μεταναστών να σέβονται και οι ίδιοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών τους για παράδειγμα. Καθώς επίσης και τα δικαιώματα τα οποία σέβεται η κοινωνία στην οποία ζουν. Δεν αποτελεί αυτό το τμήμα ένταξης. Επίσης ας λάβουμε υπόψη ότι η εμβέλεια του φαινομένου ε, ε ε, δημιουργεί το φαινόμενο, η εμβέλεια μάλλον του φαινομένου δημιουργεί την κατάσταση, ε, μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία των μεταναστών είναι εκτός Ευρώπης. Ε, αυτό δημιουργεί σημαντικότερα προβλήματα ένταξης, διότι πρόκειται για κουλτούρες πολύ μακρινές. 26 εκατομμύρια είναι άνεργοι στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Δεν είστε υπέρ του να δυσχερανθεί η μετανάστευση για ανθρώπους οι οποίοι ε, δεν θα βρουν δουλειά, δεν έχουν δυνατότητα να βρουν δουλειά στην Ευρώπη και θα φορτώσουν απλώς το κοινωνικό μας σύστημα. Δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε αυτή τη μετανάστευση. Λοιπόν κυρία Υπουργέ, όλοι είδαμε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει κυρία Υπουργέ, κυρία Κένγκελ σας ευχαριστούμε που να κάνετε ό,τι μπορείτε για να συνοψίσετε ε, στο χρόνο που έχετε τις απαντήσεις που απαιτούνται στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Σας ευχαριστούμε εκ νέου που ήρθατε και που ήσασταν έτοιμοι να αποδεχτείτε αυτήν την ανταλλαγή να Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση ε, που ήταν έντονη, ζωηρή και σίγουρα ξυπνάει σε μένα το κομμάτι αυτό που ξεπερνά ε, τα θεσμικά όργανα, το πάθος που μου οδήγησε στην πολιτική. Ένα τμήμα του πρώτου ερωτήματος. Αν είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική ένταξη. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική ένταξη όταν υπάρχουν άτομα που γεννώνται στην επικράτεια, μεγαλώνουν στην επικράτεια και δεν καταφέρνουν να ενταχθούν στον ιστό. Σε αυτή την ερώτηση πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε και ένα προβληματισμό και σε επίπεδο τοπικών θεσμών και εθνικών θεσμών. Πολύ συχνά τα άτομα όταν μετακινούνται από ένα χώρο σε άλλο έχουν ένα μεταστευτικό σχέδιο όπως αποκαλείται, ένα πρόγραμμα μεταστευτικό που δεν είναι το ίδιο σε όλες τις ομάδες ατόμων που μετακινούνται. Δηλαδή θα πρέπει να λυθεί προσεκτικά για να δοθεί μια λύση προσαρμοσμένη στο μεταστευτικό φαινόμενο. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι εκείνο της απαρχής της ένταξης. Υπάρχει και άλλο τμήμα που αφορά την εγκατάσταση, την ένταξη στην επικράτεια, στην περιφέρεια. Αυτό αφορά τις πολιτικές μιας χώρας, όσον αφορά τη στέγαση. Θεωρώ πολύ σημαντικό την πολιτική για τη στέγαση. Δηλαδή να μπορεί να ξεκινήσει κανείς Α, μια δυνατότητα ανάμειξη να συνηθίσει το άτομο. Να μην δημιουργηθούν κάποια κέντρα που να γίνονται στεία ατόμων που κλείνονται στην κοινότητά τους και δύσκολα βγαίνουν από αυτή την κοινότητα, από αυτόν τον κύκλο στον οποίο έχουν εγκλειστεί. Και αυτή είναι μία από τις πιο μεγάλες δυσκολίες που αφορούν δεύτερη και τρίτη γενιά που βρίσκονται σε γκέτο, σε αυτά τα κέντρα, όπου δεν μπορούν να έχουν επαφή με, άλλα, με άλλους ανθρώπους. Και όταν επιστρέφουν σε αυτά τα γκέτο, πολύ συχνά, εντός αυτών των κέντρων, αυτών των θυλάκων, δεν υπάρχει προστασία, διότι αφήνονται στη μοίρα τους. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις πολιτικές συγκέντρωσης των ανθρώπων στην κοινότητά τους. Να ασκήσουμε μια πολιτική διάδρασης, ανάμειξης όσον αφορά την πολιτική της στέγασης, ανάμειξης. Πολιτισμό, σχολείο. Εγώ αναφέρθηκα εκτενώ στο σχολείο στην παρέμβασή μου. Η πολιτική ένταξη βέβαια ξεκινά από τα θρανία. Στη διδασκαλία, στο σχολείο ε, θα πρέπει να ενταχθεί η μετανάστευση. Είναι κάτι εγκάσιο, δεν αφορά μόνο ένα τομέα, είναι κάτι που αφορά πολλού τομεί. Σχολείο, υγεία, Κοινωνικέ πτυχές πρέπει στο σχολείο να δημιουργηθεί και μια νοοτροπία ισότητας, ίσων δικαιωμάτων. Μέσα από το σχολείο πρέπει να μελετηθεί και η ιστορία άλλων λαών, άλλων ανθρώπων, των χωρών προέλευσης πολλών ανθρώπων. Αυτό βοηθά και διευκολύνει την επικοινωνία. Δημιουργεί φιλίες στο σχολείο. Να χρησιμοποιήσουμε και τις πολιτικές του αθλητισμού στον αθλητισμό, ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράγον ενωτικός. Ενώνει τους νέους ο αθλητισμός. Πρέπει να επενδύσουμε στους νέους για να ξεκινήσουμε την ένταξη από όταν είναι νέοι άνθρωποι, από τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης. Όταν μιλάμε για ένταξη πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλούς παράγοντες, πολλούς τομείς, να συναθριστούν όλοι αυτοί οι φορείς. Σήμερα που ξεκινά να αποκαλύπτεται το θέμα της ένταξης και το ανακαλύπτουμε, αντιμετωπίζεται σε ένα θέμα ξεχωριστό. Κανονικά το θέμα της ένταξης θα πρέπει να ειδωθεί σαν ο συνδετικός ιστός, θεμελιώδες σημείο όλων των πολιτικών και να ενταχθεί σε όλους τους τομείς. Για να ξεπεράσουμε το θέμα της ένταξης και των κοινοτήτων που δεν θέλουν να ενταχθούν, πρέπει κάθε χώρα να το εξετάσει αυτό, προσπαθώντας να δει ποιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί. Να εξεταστούν όλοι οι τομείς και από εκεί να γίνουν ιδέουσες αλλαγές για να δοθεί δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να συμμετάσχει πλήρως με πολιτικό τρόπο, με οικονομικό τρόπο στην πολιτισμική αλλαγή που μπορεί να γίνει και μέσα από το σχολείο. Μετά υπήρξε άλλο σημείο του κανονισμού του Δουβλίνου. Ο κανονισμός του Δουβλίνου μιλώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συζητήθηκε ο κανονισμός του Δουβλίνου. Πράγματι, υπάρχουν πολλά προβλήματα για πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, κατεπίγουσες ανάγκες όταν εμφανίζονται. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε να μιλούμε για κατεπίγουσες ανάγκες. Όταν βλέπω το πρόβλημα της Λαμπεντούσα, που εδώ και 10 χρόνια υπάρχει, αυτό σημαίνει να το ξεπεράσουμε να έχουμε πολιτισμό, ξεπεράσουμε τον επίγοντα χαρακτήρα του προβλήματο. Να έχουμε πολιτική πρόληψη. Πολιτική πρόληψη Δεν θα πρέπει να έχουν ευθύνη μόνο οι χώρε τη νότια Ευρώπη. Θα πρέπει να αναλάβουν ε, τι ευθύνε του και άλλε χώρε, όλη η Ευρώπη. Για να λάβει τι ευθύνε όλη η Ευρώπη, Εσεί καλείστε, εδώ σε αυτή την έδρα ακριβώ πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα, αυτή τη λειτουργία. Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια κοινότητα που εργάζεται και επεξεργάζεται όλα τα σημεία. Δεν θα πρέπει να καλείται η Ευρώπη μόνο όταν χρειάζεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι που δεν επικυρώνονται σε πολλέ χώρε. Η Ευρώπη θα πρέπει να εργαστεί σαν ενιαία κοινότητα. Εγώ θέτω το πρόβλημα. Τον επόμενο χρόνο, για τι επόμενε ευρωεκλογέ. τα επόμενα χρόνια, γιατί να μην κάνουμε μια ωραία εκστρατεία τέτοια για να προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη, το ανήκει κανείς στην Ευρώπη, να θέσουμε στις διάφορες χώρες ε, έναντι αυτής της πραγματικότητας. Το να ανήκει κανείς στην Ευρώπη τι σημαίνει. Αν δεν μπορούμε να ξυπνάμε παρά μόνο όταν είναι επίγουσα ανάγκη, είναι κάτι λάθος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σφάλματα που έγιναν κατά το παρελθόν, αλλά όχι για να κατηγορήσουμε κάποιον, να οικοδομήσουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε, να το επιδιώξουμε, να εφαρμόσουμε πρόληψη. Αυτό δεν αφορά μόνο την υποφαινόμενη σαν ε, Υπουργό Ένταξη. Εσά, σαν Ευρώπη, εσεί πρέπει να κινηθείτε, να διερωτηθείτε ποια είναι τα καθήκοντα, οι εξουσίε κάθε χώρα. Γιατί κάθε χώρα δεν κυρώνει του νόμου όταν θεσπίζονται από την Ευρώπη. Πού είναι αυτή η κοινότητα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πρέπει να ξεκινήσει ο προβληματισμό μπορούμε να κάνουμε και πολύ μεγάλη έκκληση και να ζητήσουμε βοήθεια. Αλλά αν αυτή η κοινότητα δεν έχει αυτή την έννοια της αλληλεγγύης, της ισχυρής αλληλεγγύης, το Υπουργείο Ένταξης της Ιταλίας τι να κάνει. Εμένα είναι περιθωριακό ο ρόλο μου. Οι χώρε που συμμετέχουν στην κοινότητα είναι εκείνε που πρέπει να κινηθούν για να προσπαθήσουν να προωθήσουν αυτό το μήνυμα. Εγώ απευθύνω ξανά αυτή την έκκληση. Μου το είπατε, μου το ζητήσατε, ποια είναι η θέση μου. Εγώ σα θέτω έναντι των ευθυνών σα διότι αυτό καλείστε να κάνετε εδώ πέρα. Το άλλο σημείο, όσον αφορά το αδίκημα του ε, παρανόμου μετανάστου, του κρυφού, αυτού που κρύβεται, είναι κάτι που εφαρμόστηκε στην Ιταλία. Εγώ σαν άτομο πάντα έλεγα ότι αυτό το αδίκημα δεν έχει λόγο ύπαρξης. Πιστεύω όμως ότι η Ιταλία μαζί με την Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει σαφή προβληματισμό επ' αυτού. Όχι για να πούμε ότι το αδίκημα του παρανόμου είναι αυτό που πρέπει να μπλοκάρει ε, τους παρανόμους εκεί που διακινούν τα άτομα, αλλά χρειάζονται μέσα συγκεκριμένα. Όχι που χρησιμοποιούνται σαν προπαγάνδα, συγκεκριμένα μέσα εργαλεία που όταν εφαρμόζονται, όταν υλοποιούνται αυτά τα εργαλεία να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό πρέπει να δούμε. Το συγκεκριμένο και όχι πολιτική προπαγάνδα και λόγια αυτοί που κάθεται στις, στα, στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου δεν έχουν πολιτικό χρώμα, εκπροσωπούν μια χώρα, εκπροσωπούν τους πολίτες και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται. Λοιπόν, πρέπει να θεσπίζουν εργαλεία που να προστατεύουν κάθε πολίτη ανεξάρτητος πολιτικού χρώματος. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι πολλές, προσπαθώ και εγώ να τις ομαδοποιήσω κάπως. E, uh, uh, Για το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου. Εγώ εκπλήσωμαι από αυτή την ερώτηση. Εκπλήσωμαι από αυτό το σημείο. Όταν κάνω κάποιος ασκεί πολιτική, ασκεί πολιτική διότι πρέπει να ακούσει τα μηνύματα που έρχονται από την κοινωνία. Κάποιο κάνει πολιτική και κάθεται στα έδρανα των πολιτικών αυτών οργάνων, γιατί προσπαθεί να προωθήσει πολιτικά προγράμματα. Αυτό που δεν καταφέρει να κάνει η κοινωνία, να τα κάνει αυτό πρέπει να υλοποιεί αυτά που δεν καταφέρει να κάνει η κοινωνία. Εγώ πρέπει να είμαι ταπεινά να ακούω αυτό που μου λένε οι πολίτες. Πρέπει να είμαι υπηρέτη στην υπηρεσία της χώρας μου, να ακούω τον οποιονδήποτε. Δεν έχει σημασία από ποια θρησκεία κατάγεται, ποια χώρα, τι χρώμα έχει αυτός που μου ζητάει κάτι. Πρέπει να είμαι σε θέση να τον ακούω τον άνθρωπο και να μου λέτε ότι χρησιμοποιώ τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου με εκπλήσει, διότι αυτό σκόπιμα έθεσε στο επίκεντρο το άτομο, τον άνθρωπο, στο επίκεντρο έθεσε ο Πάπας. Υπενθύμησε ότι εμείς εδώ και χρόνια δεν θυμόμαστε καν ότι αυτοί που πεθαίνουν στη Μεσόγειο είναι άνθρωποι. Στο επίκεντρο λοιπόν των πολιτικών μας, εκεί πρέπει να επιστρέψουμε, στον άνθρωπο. Αλλά δεν το λέει υποφαινόμενοι, το λέει και το Ιταλικό Σύνταγμα. Και εδώ επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα πιο ωραία συντάγματα το τελικό σύνταγμα. Μιλάει για ανθρώπου στο άρθρο 2, για το άτομο. Και πρέπει να το γνωρίζει η βουλευτή. Το άρθρο 2 του συντάγματό μα μιλά για το άτομο, το πρόσωπο, στο επίκεντρο κάθε πολιτική. Και εδώ θέτω εγώ αυτό το σημείο. Και να μου λέτε ότι εδώ κάνω χειραγώγηση αυτό που είπε, εγώ το βρίσκω παράξενο σαν ερώτηση. Διότι σαν πολιτική και σαν θεσμό πρέπει να καταλαβαίνει κανεί τα πολιτικά προγράμματα. Όσον αφορά το άλλο ερώτημα, εγώ απάντησα. Γίνεται διάλογος Υπουργού με μια Ιταλίδα βουλευτή που δεν μπορούμε να ακούσουμε. η διερμηνής είναι εκτός μικροφώνου. Έχει το λόγο η Υπουργός, η κυρία Υπουργός για να απαντήσει ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, μου ετέθηκε ένα άλλο ερώτημα που αφορά τους ανθρώπους που εισέρχονται στην Ιταλία. Λίγη ησυχία παρακαλεί ο πρόεδρος. Συνεχίζει η κυρία Υπουργό. Μιλήσατε αυτού που μπαίνουν στην Ιταλία για κάποια σύγχυση που γίνεται μεταξύ μετανάστου, παρανόμου και κρυφ... αυτού που κρύβεται. Πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει κρυφό παράνομο. Ο μετανάστης, ο λαθρέο, δεν σημαίνει ότι είναι παράνομο θέλει να διαπράξει έγκλημα, ότι φτάνει στο έδαφο μα. Ε, και ότι θέλει να διαπράξει, την είναι εγκληματία. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Αυτό βοηθά να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα και ποιε είναι οι πολιτικέ που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Πέραν αυτό, άκουσα να λέγεται ότι στη χώρα μα η νομοθεσία όσον αφορά τι ε, παναπατρισμού επιστροφέ είναι πιο ισχυρή. Εγώ είμαι υπουργό τη Ιταλία. Είμαι υπουργό ε, ένταξη τη Ιταλική Δημοκρατία. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητα της Υπουργού Ένταξης για την Ιταλική Δημοκρατία και απαντώ υπό αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, το ερώτημα που αφορούσε τις ε, επιστροφές όσον αφορά τη Δημοκρατία του Κονγκό πρέπει να τεθεί στον αρμόδιο Υπουργό της Δημοκρατίας του Κονγκό. Έχω μόνο μία επικότητα, ένα μόνο διαβατήριο. Αυτή είναι η απάντηση. Την Ιταλική, ακριβώς. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητα της Υπουργού Ένταξης της Ιταλικής Δημοκρατίας και υπό αυτή την ιδιότητα απαντώ στις ερωτήσεις. Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου που δεν ακούν οι διερμηνείς. Δεν πρόκειται περί συζητήσεως, λέει ο Πρόεδρος. Εκπροσωπεί μόνο την Ιταλική Δημοκρατία η κυρία Υπουργό, η κυρία Κέγκερ. Σαν Υπουργό τη Ιταλική Δημοκρατία, απαντώ, λέει ο κυρία Υπουργό. Αν έχετε ερωτήσει να θέσετε που αφορούν την δημοκρατία του Κονγκό, σας παρακαλώ να απευθυνθείτε προς τη ε, δημοκρατία του Κονγκό. Όσον αφορά το ότι καταγγείλατε τη 15χρονη και τους εκμεταλλευτές, υπάρχουν νόμοι, ίσως ο ρόλος ενός θεσμού είναι να μπορεί να βρει τα κατάλληλα εργαλεία, να ενισχύει τα υπάρχοντα εργαλεία, και όταν είναι αδύναμα τα εργαλεία να τα ενισχύει, τα μέσα να τα ενισχύει, ούτως ώστε να χορηγείται προστασία στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εκβιάζονται οι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν επικοδομητικές κριτικές να βοηθούν τις διοικητικές αρχές στην τοπική αυτοδίκηση για να παρέχουν τη σωστή προστασία. Λοιπόν, Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που αφορά τους ανθρώπους που καταφθάνουν. Πώς μπορούμε να σεβαστούμε τους νόμους στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι σε κάθε χώρα όταν γίνεται λόγος για πολίτες πρέπει πάντα να ξεκινούμε την προϋπόθεση ότι για κάθε πολίτη, εγώ δεν έκανα ποτέ διακρίσεις, ότι πρέπει να καθορίσουμε ως πολίτη λοιπόν οποιοδήποτε άτομο, οποιοδήποτε άνθρωπο. Το θέμα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων είναι θεμελιώδες θέμα για οποιονδήποτε. Και αν κάποιο παρανομεί υπάρχει σχετικό νόμο, υπάρχει ο νόμο γι' αυτό. Αν κάποιο διαπράττει βία η πράξη, αν, εάν υπάρχουν παραβάσει, υπάρχει ο νόμο γι' αυτό. Το βασικό θέμα είναι ότι δεν έχει χρώμα η παραβίαση, δεν έχει εθνικότητα και δεν ανήκει σε μια κοινότητα. Αλλά η βία όταν εφαρμόζεται από κάποιον ε, ε, γίνεται από αυτόν. Πρέπει να πάμε στο αίτιο και να μην προσπαθούμε να δώσουμε εθνοτικό χαρακτήρα στη βία. Ε, αυτό πρέπει να προσέξουμε. Όχι τόσο πολύ την κοινότητα όταν κάποιος διαπράττει ένα δίκημα, μια βία πράξη. Σίγουρα έχασα και πολλά άλλα σημεία, άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν μπορώ να τα καταφέρω να απαντήσω όλο και αν κάτι λησμόνησα που είναι θεμελιώδη σημασία είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, κυρία Κουίνγκε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση ε, που έλαβε χώρα. Ευχαριστούμε για το θάρρος σας, για την αποσίωσή σας. Αν ερμηνεύω πιστά τα συναισθήματα, τα ομόφωνα των μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι η πρόβλεψη και η προσδοκία ότι δεν θα είναι τελευταία φορά που θα προσκληθείτε στην Επιτροπή μας και σας απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές, καλύτερες ευχές για τις προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε ως υπουργό Ένταξης της Ιταλικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους όλων.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 Now. Κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Υπουργό και το επιτελείο της. Σίγουρα ήταν ένα φλέγον ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Καυτό. Παρακαλώ όμως, όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν ήσυχα διότι το σημείο, να σας πω, 25, το οποίο είναι και το σημαντικότερο, έχει συρρυκνωθεί από την ένταση που είχε αυτή η συζήτηση. Τώρα, το επόμενο θέμα αφορά ε, την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το πακέτο για τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε και τους δύο εισηγητές εδώ, τον κύριο Γιάνν Φιλίπ Άλμπρεχτ, για τον κανονισμό και τον κύριο Δημήτριο Δρούτσα για την οδηγία. Θα γνωρίζετε όλοι ότι αυτό το θέμα είναι κέριο και επίκαιρο και δυστυχώς ε, θα έχουμε λιγότερη ώρα για να ασχοληθούμε με αυτό στην ημερήσια διάταξη διότι ακόμα ε, έχουμε να ε, διεξάγουμε και την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης που προβλέπεται για, την... για τις 6 παρατέταρτο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο λοιπόν. Και δεδομένη της εκείνης συνεδρίασης, παρακαλώ να μην κάνουμε τους συναδέλφους να περιμένουν πάρα πολύ. Σας παρακαλώ λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το χρόνο όσο καλύτερα μπορείτε για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Προτείνω να προχωρήσουμε χωρίς καμία καθυστέρηση να ακούσουμε τους συζητητές μας και μετά να αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και συμπεριλαμβανομένων και των απόψεων της ε, Επιτροπής και του Συμβουλίου. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε για τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σίγουρα είναι απογοητευτικό ότι έχουμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε. Ε, δεν έχουμε μείνει και πολύ εξάλλου. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι σύντομος όσο γίνεται. Να σας ε, ενημερώσω με λίγα λόγια για το πού βρισκόμαστε και ύστερα ενδεχομένω θα έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και επί της ουσίας, κάτι που δεν είναι δυνατόν τώρα. Σχετικά με τη διαδικασία τώρα. Υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την ε, επίτευξη συμβιβασμών. Φυσικά παραμένει μια πρόκληση για εμάς να οδηγηθούμε σε συμβιβασμούς για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ήδη έπρεπε να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα ελπίζω να ψηφίσουμε το αργότερο τον Οκτώβριο. Επίσης τον Οκτώβριο θα συνεδριάσει και το επόμενο σχετικό συμβούλιο και ελπίζω να έχει κάποια έστω και γενική προσέγγιση, να έρθει στις διαπραγματεύσεις, στους τριμερείς διαλόγους με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ε, τώρα κοιτάζοντας τους συμβιβασμούς αλλά και την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η Ιρλανδική Προεδρία, μπορώ να πω ότι δεν απέχουμε και πολύ. Πλησιάζουμε, έχουμε την προσέγγιση που θα θέλαμε, θέλουμε να εναρμονίσουμε τους, ε, τις διατάξεις του κανονισμού που ισχύει από το 1985. Έχουμε φυσικά τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και τη μαζική χρήση προσωπικών ε, δεδομένων στις εμέρες μας, το οποίο αποτελεί πρόκληση και για τους πολίτες και για τους καταναλωτές, καθώς επίσης και για όσους ελέγχουν τα δεδομένα και την κίνησή τους. Πρέπει λοιπόν να συμφιλιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα στις συνεδριάσεις μας και Επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία με τους συζητητές είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε και να φτάσουμε σε συνένεση, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δείξουμε στους πολίτες ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να δώσουμε ένα νέο πλαίσιο στους πολίτες μας για την προστασία δεδομένων, ιδιαίτερα τώρα Ανυπομονώ λοιπόν για τις εξελίξεις και ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να έχετε εμπιστοσύνη και στους κοιόδης εισηγητές σας και σε μένα ως εισηγητή. Φυσικά χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος, αλλά πραγματικά εγώ θα ήθελα να πιέσω έτσι ώστε να επισπεύσουμε την διαδικασία και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο έτσι ώστε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ελπίζω αμέσως μετά τις θερινές διακοπές να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλμπρεχτ. Συγγνώμη για τον λίγο χρόνο που έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για την συνοπτική παρουσίαση που μας κάνατε. Τώρα σειρά έχει ο κύριος Δρούτσας για να μας παρουσιάσει την οδηγία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω το παράδειγμα του κύριου Άλμπρεχτ και θα είμαι πολύ σύντομο. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ε, ακολουθώ τα όσα είπε ο κύριος Άλμπρεχτ. Το πακέτο, για μας είναι πακέτο και οδηγία και ο κανονισμός. Τώρα, ε, όσον αφορά το τι γίνεται με την οδηγία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σας πω ότι η οδηγία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ο κανονισμός. Οι εξελίξεις είναι πιο θετικές. Καταρχάς μπορώ να πω ότι η συνεργασία με τους σκιώδεις είναι εξαιρετική. Και εδώ να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για την ε, ανοιχτόμυαλη προσέγγιση που έδειξαν και τη συνεργασία τους και έπειτα να πω ότι προσπαθήσαμε, ότι προσπαθώντας μάλλον να οδηγηθούμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες καταφέραμε πάρα πολλά και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στην οδηγία υπάρχουν δύο διαφορετικές σε τρόπον την κατηγορίες άρθρων. Στις ε, προηγούμενες συζητήσεις μας, αν θυμάστε, ο στόχος της οδηγίας ήταν να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο εναρμονισμένη γλώσσα με τον κανονισμό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά άρθρα στην οδηγία τα οποία ε, είναι παρόμοια με αυτά του κανονισμού. Αυτό που εμείς κάνουμε τώρα είναι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό, πώς θα διατυπωθούν αυτά τα άρθρα και να τα πάρουμε έτσι αυτούσια και να τα εισάγαγουμε στην οδηγία. Κατά τα άλλα, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, όπως είπα. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι μετά από μία-δύο το πολύ συναντήσεις και οδών εισηγητών θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για την οδηγία. Πρόεδρε, ας, τελειώ, ας με αφήσετε να τελειώσω τώρα με λίγα λόγια για την προσέγγιση την συνολική, ως πακέτο. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία εποχή νέα, μία εποχή μετά το πρόγραμμα PRISM στην Ευρώπη. Πραγματικά αυτό ήταν αφύπνιση η κοινή γνώμη είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη όσον αφορά την προστασία δεδομένων και πιστεύω πως ως Κοινοβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε αυτές τις ανησυχίες και τις ευαισθησίες τα σοβαρά στη δουλειά μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις εργασίες μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Γιάννη πιο πριν. Και όσον αφορά την οδηγία λοιπόν, να επαναλάβω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο τουλάχιστον πρέπει να επιμείνουμε για την προσέγγιση ως σύνολο, ως πακέτο, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει την ίδια με να απολαμβάνει τις ίδιες μεταχείρισεις με τον δημόσιο τομέα. Γι' αυτό λοιπόν και είναι σημαντική η προσέγγιση ως πακέτο, ως σύνολο. Κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους, σε όλες τις πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο να μην εγκαταλείψουν την ε, προσέγγιση αυτή και να επιμείνουν στην αρχική προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι εμεί το Κοινοβούλιο ήμασταν εκείνοι που είπαμε ότι θέλουμε μία ενιαία νομοθετική πράξη που θα καλύπτει όλους τους τομείς ε, ε, της προστασίας δεδομένων. Ας τιμήσουμε λοιπόν την ε, υπόσχεσή μας αυτή, ας στηρίσουμε την προσέγγιση ως σύνολο και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν και να το ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δρούτσα. Κύριε Φώση, είστε σχεώδης εισηγητής. Έχετε το λόγο. Κρατήστε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και εγώ να είμαι πάρα πολύ σύντομο, γιατί ξέρω πω δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω και του δύο εισηγητέ για την δουλειά που έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε εντατικότατα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και μάλιστα τώρα, λίγο πριν τις θερινές διακοπές, φαίνεται Ηράκλειο έργο. Εμείς ελπίζω, ελπίζω Εύχομαι τον Οκτώβριο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Βέβαια, μόλις γυρίσουμε το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε. Έχουμε όμως τον Οκτώβριο κατά νου, αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζω πως και οι δύο εισηγητές βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Τώρα, επί του περιεχομένου, πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να σας ε, αναφέρω τις λεπτομέρειες μια που δεν υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό πιστεύω είναι συλληνετό απλά να πω ότι θα περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο, στο μεταξύ θα εργαζόμαστε να θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα όσον αφορά αυτά που μας είπε μόλις ο κύριος Δρούτσας για την οδηγία, όντως πρέπει να αναλογιστούμε εάν στην οδηγία ακολουθούμε τη σωστή οδό, εάν θα έπρεπε μήπως να ήμασταν πιο ε, γενική, να έχουμε πιο ευρύ πεδίο δράση. Σε γενικέ γραμμέ όμω πιστεύω ότι είμαστε πολύ ε, ευχαριστημένοι. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο με αυτήν την προσέγγιση ω πακέτο και ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, να πω ότι ε, επιθυμούμε τι υψηλές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων αλλά και σαφή και λειτουργική νομοθεσία. Δεδομένου ότι πρόκειται για ο κανονισμός τουλάχιστον για ένα κείμενο άμεσης εφαρμογής ε, ο νομοθέτης ε, έχει καθήκον να συμφωνήσει σε μια διατύπωση που θα είναι ψηλής ποιότητας και ξεκάθαρη. Ε, από όταν έγινε προσωρινή Γη ηγήτρια σε δύσκολες στιγμές για την ομάδα μας μετά το ατύχημα του κ. Άλβαρο προσπάθησα επανειλημμένως ε, να εντοπίσω και να προσδιορίσω το ακριβές νόημα τόσο του κειμένου της Επιτροπής όσο και ορισμένων τροπολογιών του εισηγητή και άλλων. Χαίρομαι που ο εισηγητής ε, δέχτηκε ορισμένες από τις ε, προτάσεις ε, τροπολογιών της ομάδας μας. Νομίζω ότι έτσι διευκρινίζονται τα πράγματα. Επιθυμώ τις καλύτερες σχέσεις με την υπόλοιπη ομάδα Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε προγραμματίσει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Να πω στο Γιάννη ότι δεν είμαι σίγουρη πως θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συνένεση. Ε, ίσως γιατί η συνένεση θα σήμαινε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή αντί για το μέγιστο. Ορισμένες ιδέες που θα εξασφάλιζαν συνένεση ενδεχομένως ε, δεν θα εξυπηρετούσαν το συμφέρον των πολιτών. Είναι σημαντικό να μην κάνουμε πλούσιους τους δικηγόρους απλώς. Ακόμα και πριν το, τις αποκαλύψεις για το πρίσμε, γνωρίζαμε ένα μεγάλο κομμάτι της πραγματικότητας και χρωστάμε στους πολίτες μας ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, με την επανσογή της ρήτρα την οποία φέρεσε η Επιτροπός Ρέντινγκ και η βοηθή της και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μυστικέ υπηρεσίε θα δίνουν λογαριασμό είτε μέσω της οδηγίας είτε μέσω του κανονισμού είτε μέσω πολιτικών ή διπλωματικών οδών. Εγώ είμαι πρόθυμη να βοηθήσω προκειμένου το κείμενο να μας κάνει περήφανους. Και να είναι εύκολα εφαρμόσιμο. Thank you. Κύριε ευχαριστώ πολύ. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ε, εισηγητές. Είναι μια πολύ πλοκή δουλειά, ηράκλειο έργο. Συζητούμε πάρα πολύ καιρό και φυσικά πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιον συμβιβασμό. Βέβαια, οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες που έχουμε. Περιμένουν ε, πραγματικά πάρα πολλοί από εμά όταν λένε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το, το έργο μας μέσα σε αυτή την νομοθετική περίοδο, δυστυχώς δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε άλλο. Συζητάμε εδώ και ένα χρόνο για αυτό το θέμα, σε αυτό το στάδιο και έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Και όλες αυτές οι συζητήσεις επί συζητήσεων πρέπει να οδηγήσουν κάπου. Δεν θα επεκταθώ όμω σε αυτό. Σε γενικέ γραμμέ θα ήθελα να πω ότι έχουμε επίση ευθύνη να φέρνουμε όχι μόνο ποιότητα, αλλά να το κάνουμε αυτό και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που ήθελα να πω, η προσέγγιση ως πακέτο ήταν ένας μεγάλος αγώνας και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Προβλέπετε σφαγή και σας το λέω αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά την προσέγγιση ε, μαζί με τον ε, κανονισμό, όμως ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι μία ευχή. Ελπίζω, λοιπόν, και είναι κάτι που το λέμε και εδώ και πολύ καιρό, όπως και στις υπόλοιπες επιτροπές, έτσι και σε αυτήν εδώ την επιτροπή, να έχουμε επιτέλους μία ή δύο ώρες στη διάθεσή μας, όταν θα έχουμε όλους τους συμβιβασμούς ε, μπροστά μας, να μπορέσουμε να τους συζητήσουμε, να τους εξηγήσουμε και όχι σε κλειστό κύκλο, αλλά να είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε το κοινό όλους το τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, να πω πως εύχομαι πραγματικά να υπάρξει ευρία κατανόηση και συνένεση και πραγματικά να επαναλάβω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο στην Επιτροπή, αλλά πρέπει να βρούμε χρόνο και γι' αυτό το ε, θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάιντεν είναι μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι εργασίες να ολοκληρωθούν και να ψηφίσουμε σύντομα διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα με, το, με τις αποκαλύψεις για το πρόγραμμα PRISM και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε και είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και να διαπραγματευτούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα ε, το άρθρο 42 της ε, αρχικής ε, εκδοχής του κειμένου της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να επαναχρησιμοποιήσουμε λοιπόν το άρθρο 42. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι πεπισμένος ότι ο κύριος Άλμπρεχτ και οι σκιώδες εισηγητές του εργάζονται σκληρότατα για τις συμβαστικές τροπολογίες. Όμως, ως ε, μέλος αυτής της ε, Επιτροπής να πω ότι είμαι ανυπόμονος. Πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Τώρα μας λέτε ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή τον Οκτώβριο και θέλω να ρωτήσω, μας το εγγυάσει αυτό ο Γιάνν Φίλιπ. Διότι εμείς ως ε, μέλη της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς θέλουμε να τη συνεχίσουμε αυτή την εσωτερική αγορά. Και πραγματικά χρειαζόμαστε μία πλήρη προσέγγιση, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έρχονται εκλογές. Και αν το Συμβούλιο καθυστερήσει, εμείς θα οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα μετά τις ευρωεκλογές. Και αυτό θα μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Και φυσικά καταλαβαίνω απόλυτα ότι ένα συμβάν όπως υποκαλύψεις για το πρίσμα μας δίνει πρόσθετο φόρτο εργασίας, αλλά αν τα πάρουμε όλα αυτά μαζί μας στις επόμενες εκλογές δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δώστε μας λοιπόν σας παρακαλώ αποτελέσματα και γρήγορα. Και την επόμενη φορά θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ κύριε Βάντεκαμ. Κύριε Κυρία Ρομέρο χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς η ομιλήτρια. Πράγματι, οι γερμανικές εκλογές επηρεάζουν το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο όμως. Η Λιθουανική Προεδρία είπε σήμερα πως θα χειριστεί το θέμα της προστασίας των δεδομένων ως πακέτο, τον κανονισμό και την οδηγία μαζί. Όμως στο Συμβούλιο ε, έχει εμφανιστεί ένα μπλοκάρισμα. Οπότε σε τι οφείλεται αυτό το μπλοκάρισμα. Οφείλεται στην ε, συμπρίληψη του δημόσιου τομέα, σε κάποιο άλλο θέμα. Δεν ξέρω πότε ε, ε δεν ξέρω αν έχει, ξέρει η, η, η για αυτό το θέμα. Ε, πώς θα λυθεί το ζήτημα αυτό. Ε, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το θέμα του κανονισμού. Ε, σίγουρα αν προχωρήσουμε στον κανονισμό είναι σημαντικό, αλλά τώρα έχουμε με το πρίσμ και το μεγάλο ζήτημα της εξοεδαφικότητας. Γιατί ακόμα και με μια ευρωπαϊκή οδηγία πάλι δεν έχουμε ασφάλεια. Μακάρι να διαθέτουμε μια οδηγία το συντομότερο δυνατό. Τι γίνεται όμως με την εξοεδαφικότητα. Η, ο πατριωτικός νόμος και όλοι οι άλλοι νόμοι που ψηφίζουν στις ΗΠΑ ε, είναι νόμοι που κατ' εξαίρεση εφαρμόζονται εκτός της, ε, Ευρωπαϊκής, εκτός της, ε, του, των, ε, της των ΗΠΑ επιτρέπουν μυστικές φυλακές, επιτρέπουν πολλά πράγματα Οπότε, ποια είναι η δική μας θέση. Θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε όλες τις απαντήσεις με το πακέτο προστασίας των δεδομένων, παρόλο που και αυτό έχει προβλήματα. Sorry, we so Ε, πρόεδρος, έχουμε καθυστερήσει δυστυχώς. Είμαι σίγουρος όμως ότι ε, το θέμα αυτό θα μείνει στην ατζέντα. Αμέσως μετά την στερινές διακοπές θα επιστρέψουμε. Ο χρόνος όμως πιέζει. Θα δώσω ένα λεπτό στην Κομισιόν και μετά στους συζητητές. Θέλει όμως η Κομισιόν να κάνει κάποια σχόλια. Ένα λεπτάκι παρακαλώ μόνο, όχι παραπάνω. Και το Συμβούλιο βέβαια. Ε, από πλευράς Κομισιόν να πω ότι καλωσορίζουμε την σκληρή δουλειά στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό το πακέτο να υιοθετηθεί σύντομα, γρήγορα. Ε, είμαστε υπέρ του χειρισμού του ως πακέτου και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο θέλει να καταλήξει σε υιοθέτηση τη εκθεση του μέσα στην, να εκθεθεί μάλλον το πακέτο ε, με, κατά τη διάρκεια του. Το Συμβούλιο. Όπως είπε και ο Υπουργός πριν από λίγο, το πακέτο αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Θα εργαστούμε σκληρά στο Συμβούλιο για να πετύχουμε πρόοδο. Η προσέγγιση μας θα είναι προσέγγιση πακέτ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια πιο πολύ αρχικά με τον κανονισμό, αλλά θα συνεχίσουμε παράλληλα τις συζητήσεις και για την οδηγία. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση κυρίας Ρομέρο Λόπες, δεν έχει ληφθεί απόφαση από το από το Συμβούλιο για το πεδίο εφαρμογή των δύο αυτών εργαλείων νομικών κειμένων. Αυτό θα συζητηθεί αργότερα. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση αυτή τη στιγμή για το πεδίο εφαρμογή. Ωραία. Και πάλι ο λόγος στους ηγητές. Επιμένω, το θέμα αυτό θα ξανασυζητηθεί μετά τις θερινές διακοπές, μετά το καλοκαίρι. Ε, σας δίνω το λόγο προκειμένου να ξεκινήσει μετά η κοινή συνεδρίαση ε, των δύο επιτροπών μας. Ευχαριστώ, κ. Σάλμπρεκτ. Ε, ευχαριστώ πολύ και τους ε, σκιώδης που φέρουν μεγάλο βάρος και αυτοί. Οι συναντήσεις μας είναι πολλές και αρκετά περίπλοκες θα έλεγα. Ορισμένες ομάδες ε, παραπονέθηκαν για το μεγάλο αριθμό των συναντήσεων. Ε, βάρος φέρει και η γραμματεία. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, συνενετικής προσέγγισης, συμφωνώ ότι τελικά δεν πρόκειται όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι με ένα τέτοιο κανονισμό που άπτεται τόσων διαφορετικών τομέων, έχει τόσες διαφορετικές πτυχές, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Ο στόχος ιδανικά είναι να έχουμε κοινού κανόνες. Και εδώ στο Κοινοβούλιο συμφωνούμε λίγο πολύ, συμφωνήσαμε λίγο ως πολύ για το ψήφισμα του 2011, όπου αναφερόμασταν σε ενιαίο σε ενιαίους κανόνες ε, που θα ξεκινάνε από το επίπεδο προστασίας της οδηγίας του 95. Τώρα, άμα δούμε και ορισμένε από τις τροπολογίες που έχετε προτείνει εσεί, ε, πολλές από αυτέ είναι κάτω από τον πύχη της οδηγίας του 95. Οπότε δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτό που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Θα πρέπει όλοι μας κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Η... Στις δικές μου προτάσεις προσπαθώ να λάβω υπόψη πολλές ανησυχίες, πολλές επιφυλάξεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να λάβω υπόψη τα πάντα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα κανονισμό που θα γίνει δεκτός από ένα μεγάλο αριθμό μελών, δεν θα ήταν σωστό να ε, υποχωρήσουμε σε σχέση με αυτό που έχουμε αποφασίσει στο παρελθόν. Οι πολίτες θέλουν να είμαστε ενωμένοι, ιδιαίτερα στις συζητήσεις μας για το Κοινοβούλιο. Ε, συγγνώμη, στις μας με το Συμβούλιο. Ο κ. Δρούτσας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες μας, τη γραμματεία, τις πολιτικές ομάδες πάρα πολλές ε, ώρες σκληρής δουλειάς και γι' αυτό τους εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας, λέει ο Πρόεδρος. Είναι ουσιαστικό το θέμα. Θα το παρακολουθήσουμε και συνεχίζουμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι φεύγουν, παρακαλώ πολύ, με ησυχία. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, για τη συνεργασία σας. Τελευταίο θέμα. Ζητάμε συγγνώμη από τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ που καθυστερήσαμε. Πέσαμε λίγο έξω στο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Ζητούμε συγγνώμη. Σημείο 25. Ανακοίνωση Επιτροπή σχετικά με την μεγιστοποίηση της, ε, των αναπτυξιακών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Ε, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Θεμάτων, ο κ. Ζόζεμπεργκ, μέρος της Κομισιόν, εκεί, στο βάθος, και ο εκπρόσωπος της, η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ, η κυρία Ελένη είναι επίσης εδώ. Μετά θα δώσουμε λόγο στον, το λόγο στον κύριο Hemingway. Ε, και θα περάσουμε στα μέλη. Καταρχήν όμως λόγος στην κυρία Κρέτου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ, για ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων εν ώψη του διαλόγου υψηλού επίπεδου για τη διεθνή μετανάστευση που θα λάβει η χώρα τον Οκτώβριο του 2013 στα κεντρικά του, του Εθνών. Ιδιαίτερα σε μια εποχή κοινωνικονομικής αστάθειας ε, οδηγούμαστε σε προβληματισμό. Η οικονομική κατάσταση, η ανεργία, η ανασφάλεια σε τοπικές κοινωνίες οδήγησαν σε αύξηση της φτώχειας και ε, στερήσει σε, όλ, όλο τον κόσμο. Η μετανάστευση πολλές φορές είναι μοναδική λύση που βρίσκουν κάποιοι για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή ζωή και όρους εργασίας. Για την Ευρώπη που αντιμετωπίζει κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, με τον ενεργό πληθυσμό να μειώνεται και τον αριθμό των ατόμων που εξαρτώνται να αυξάνεται, η μετανάστευση δεν είναι η μόνη λύση, αλλά πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της κοινή λύσης. Ε, η νόμιμη και ελεγχόμενη μετανάστευση δίνει λύσεις και για τη χώρα πλεύση και για τη χώρα προορισμού. Ε, τα εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες ε, χρηματοδοτούν τις τοπικές κοινωνίες αλλά και από την άλλη πλευρά οι μετανάστες ε, πληρούν θέσεις ε, εργασίας τις οποίες οι ντόπιοι δεν θέλουν να ε, εκμεταλλευτούν. Το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βελτιώσει το ρόλο που παίζει η μετανάστευση με έναν τρόπο συντονισμένο και συνεπή. Χαίρομαι που η Κομισιόν έχει την ίδια προσέγγιση. Ιδιαίτερα εκτιμώ την ειδική αναφορά στη γυναίκα, στα παιδιά και τις ε, πολιτικές ε, ε, κατά της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Της διακίνησης ανθρώπων. Θα πρέπει να εστιαστούμε στα εξή. Από την πλευρά της Επιτροπής μας τουλάχιστον. Δεδομένης Δεδομένου ότι ο κόσμος είναι αλλοεξαρτάται αυτή τη στιγμή και ότι η φτώχεια είναι ε, διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό ε, ε, να ρυθμίσουμε τη μετανάστευση. Οι διαδικασίε λήψη αποφάσεων στο Βορρά και στο Νότο θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των φτωχότερων ανθρώπων και να μην πλήττουν ε, τι προοπτικέ ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σύνδεσμο ανάμεσα στην μετανάστευση και την ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ατζέντα μετά το 2015. Η Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Δημογραφία μετά το 2014 ε, κατέληξε σε, μια, σε ένα κείμενο το οποίο δίνει ε, συστάσεις ε, για, μάλλον, ε, στο οποίο αποδεικνύει τις ε, ευκαιρίες που δημιουργούνται από την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Δεύτερο θέμα είναι η βελτίωση των θετικών πτυχών της μετανάστευσης μεταξύ χωρών του Νότου. Ανάμεσα δηλαδή σε χώρες που αντισόμενες χώρες. Ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως αυτό το φαινόμενο, διότι σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο, ε, οι πηγές μάλλον, τα δεδομένα είναι ελλειπή. Ίσως αυτή η μετανάστευση είναι αποτελεί το 47% του συνολικής μετανάστευσης από χώρες του Νότου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διευρύνουμε την δράση μας και στο πλαίσιο της μετανάστευσης μεταξύ χωρών του Νότου. Για παράδειγμα, διευκόλυνση ε, των εμβασμάτων μεταξύ τέτοιων χωρών διότι όπου επιτρέπονται συνήθως τα εμβάσματα αυτά είναι υψηλότερα από, αυτά, από τις χώρες του Βορρά προς τις χώρες του Νότου. Διότι στο, στις χώρες του Βορρά για παράδειγμα είναι πιο ακριβέα τέτοιου είδους εμβάσματα. Τέλος, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική δεν υποσκάπτεται αλλά αντιθέτως ε, υποστηρίζεται από άλλες πολιτικές. Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχουν 32, εκατομμύρια μετανάστες με αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση στα νότια σύνορα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βελτιώσουμε το σεβασμό της αξιοπρέπειας αυτών των μεταναστών που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των ε, ε, αναγκών σε εργατικό δυναμικό. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε την κινητικότητα ε, εργαζομένων με προσόντα, μεταναστών με προσόντα εκεί όπου χρειάζεται και να ε, βελτιώσουμε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να κατάφερα να προσδιορίσω τα καλύτερα μέτρα για την βελτίωση του ρόλου των μεταναστών ε, σε συντονισμό με τη, με σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα διεθνή όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρήτου, τώρα θα προχωρήσουμε αμέσω με την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, με την Γαμαδελταχούμ, κύριε Ρόσενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Συνεπρόεδρο που τόνισε αυτά τα ζητήματα, ζητήματα τα οποία μας ανέπνευσαν για να σχεδιάσουμε αυτήν την Ανακοίνωση. Η ανακοίνωση εγκρίθηκε στις 21 ε, Μαΐου πριν από 6 εβδομάδες. Ε, συντάχθηκε από κοινού με την ε, ΓΔΚΟΜ και την ΝΤΕΦΚΟ και εγκρίθηκε από τον, τους επιτρόπους και Μάλιμστρομ. Ο σκοπός της ανακοίνωσης είναι διτός. Καταρχάς στοχεύει να προετοιμάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στα στον επικείμενο διάλογο στην Νέα ΕΕ τον Οκτώβριο, διότι εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με μία φωνή και θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να το επιτύχουν αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η πρόθεσή μας, ξεκάθαρη, και, ξεκάθαρη ε, πρόθεση και δεύτερον θα δείτε ότι η δομή είναι ίδια με τους ε, γύρους τρογγυλής τραπέζης, ιδιαίτερα τα σημεία 2 έως 5. Επίσης υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος της ανακοίνωσής μας, τον οποίο θα βρείτε στην, ε, στο τμήμα 6. Πάμε λίγο πέρα από τον εαυτό μας, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για να μπορέσουμε να εντάξουμε τους στόχους της μετανάστευσης και να, συνδε... να τους συνδέσουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι το κάνουμε τώρα. Τώρα θα σας αναφέρω και τον τρίτο στόχο που έχουμε. Ήταν ένας κρυμμένος στόχος τροποντινά και θέλει να δείξει λοιπόν ο στόχος αυτός την εμπειρία που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε επιτύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν πρωτοπόροι μια ε, εξωτερική μεταναστευτική πολιτική με τέσσερι πυλώνε συμπεριλαμβανομένου τη ε, μεταναστευτική ανάπτυξη και αυτό ήταν κάτι που ενέπνευσε διάλογο όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω και εκτό στα πλαίσια της μεταναστευτικής σταθερότητας όπως ονομάστηκε. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που ανέπτυξαν αυτούς τους συνδέσμους ανάμεσα στην μετανάστευση και στην ανάπτυξη με λεπτομερή τρόπο και να σας πω ότι εμπνευστήκαμε από τα από τα κόνσεπτ για τα PCD που προήλθαν μάλιστα από το Κοινοβούλιο εδώ στη δεκαετία του 90 και αυτό λοιπόν ενέπνευσε εμάς την δουλειά της Επιτροπής εδώ και 15 χρόνια και πιστεύω πως αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα και φαίνεται και από την ανακοίνωση. Και επίσης πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτόν τον κοινό χώρο ελεύθερης μετακίνησης, το Σέγγεν δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανους και έτοιμους να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τη γνώση μας με άλλους εταίρους στον κόσμο έτσι ώστε να βελτιώσουμε τους, ε, και να αναρμονίσουμε τους στόχους για τη μετανάστευση. Τώρα όσον αφορά την ε, ανακοίνωση, όπως σας είπα, η δομή της ε, ακολουθεί τη δομή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης και φυσικά εκεί αναφερόμαστε στην, αναπτυσσόμενη κοινότητα και λέμε πως αν πρέπει αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τον 21ο αιώνα, πρέπει να ε, εντάξουμε πλήρως το ρόλο τη μετανάστευση και τη κινητικότητας ε, και αυτό πρέπει να είναι κύριος στόχος μας. Πρέπει να ε, πιάσουμε το δυναμικό, να χαλιναγωγήσουμε το δυναμικό που έχει αυτό και να το μοιράσουμε ανάμεσα στις ε, χώρες με διαφορετικά επίπεδα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει όχι μόνο χάραξη πολιτικής, πρέπει να δούμε και πέρα από τους ε, παραδοσιακούς τομείς, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τη διαρροή εγκεφάλων, επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, ενδοκινοτική μετανάστευση, με την μετανάστευση από νότιες χώρες σε νότιες χώρες, από αναπτυσσόμενες σε αναπτυχωσόμενες, με την κινητικότητα, να μην εστιάσουμε μόνο στην ε, μετανάστευση αλλά και στην κινητικότητα και τις ε, σύντομες ε, αποστάσεις κινητικότητας, να δούμε τι γίνεται με την αστικοποίηση και με την μεγαλύτερη σροή μετανάστευσης και φυσικά με την κλιματική αλλαγή και το πώς μπορούμε να εντάξουμε και να ερμηνεύσουμε την μετανάστευση στα πλαίσια αυτής. Γενικά τώρα το μήνυμα της εκκινητικότητας στη μετανάστευση πρέπει να είναι ότι διευκολύνει την ένταξη και την προσαρμογή και αυτό στα πλαίσια των στόχων μετά το 2015. Επίσης, ε, ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, με τη διακίνηση, με το λαθρεμπόριο. Εδώ τονίζουμε ότι τα δικαιώματα των μεταναστών και η προάσπιση τους ε, είναι κάτι το οποίο ήδη αντιμετωπίζουμε ε, σε ένα διεθνές νομικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο εμείς θεωρούμε επαρκές. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για καλύτερη εφαρμογή αυτών που έχουν συμφωνηθεί και να επιβάλλουμε την προστασία των ε, δικαιωμάτων των ε, μεταναστών, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, τώρα, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. επίτηδες δεν μιλάμε για ε, όργανα και συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός ε, στο πρωτόκολλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών και την πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Επίσης, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης νούμερο 3 έχει να κάνει με την συνεργασία, με τις εταιρικές σχέσεις και με την ε, αποτελεσματική ένταξη των μετανάστευση της μετανάστευσης στις υπάρχουσες ε, πολιτικές. Εδώ πέρα αντιλούμε από την εμπειρία μας από τους ε, διαλόγους και τις διάφορες μεθόδους που έχουμε ακολουθήσει. Επίσης γίνεται λόγος για πολυμερή συνεκτικότητα στη μετανάστευση και στα πλαίσια αυτά να πω ότι την, αναγνωρίζουμε την αξία του Παγκόσμιου Μεταναστευτικού Φόρουμ, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα, στους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς και όχι μόνο. Επίσης, καλωσορίζουμε τον ε, IOM ως τον ε, ηγετικό οργανισμό στον τομέα αυτό και ζητούμε να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και να είναι προορατικός και επίσης αναγνωρίζουμε και το έργο του Γενικού Γραμματέα της ΑΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ανάπτυξης του κύριου Πίτερ Σάτερλαντ, ο οποίο επίσης έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτικών αυτών. Τώρα, κύκλο στρογγυλής τραπέζης 4, κινητικότητα και επιπτώσεις της κινητικότητας στην ανάπτυξη εδώ ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα υφιστάμενα εμπόδια που υπάρχουν ε, για, να την ε, κινητικότητα και να έρθουν τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα που, είναι... που εμποδίζουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Επίσης, για να προωθήσουμε τις επιπτώσεις, ε, τον αντίκτυπο της μετανάστευσης και της κινητικότητας, θεωρήσαμε καλύτερο να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση και την νομοθεσία στην, ε, όσον αφορά το, μεταναστευτικό ε, δίκαιο και την ε, εργασία. Και επίσης αναγνωρίσαμε ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις ε, ε, το έργο μας όσον αφορά την απόκτηση ε, προσόντων και δεξιοτήτων, τα δικαιώματα συνταξιοδότησης ή δυνατόν σε διεθνές επίπεδο. Αυτά προς το παρόν ε, εν για τους γύρους στρογγυλής τραπέζης. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά θέματα και προσπάθησα να είμαι πλήρης. Ο συνάδελφός μου από τη ΔΕΛΤΑΧΟΜ θα σας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόζενμπεργκ. Παρακαλώ όλη μέρα ζητούσα από τους συναδέλφους να είναι σύντομη. και τώρα σχεδόν μας τελειώνει ο χρόνος διερμηνίας, οπότε σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας αυτό έτσι ώστε να έχουμε κάποιο χρόνο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ανοίγω τώρα ε, τον... Ε, μάλλον πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπουργκάντ από την Δέλτα Ντεύκο. Έχετε το λόγο. Thank you. Yes. Okay, I will shift to French. I see that I have the luxe of having interpreters. Um, bien. Eh bien, nous Καλώς εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος την διοργάνωση αυτής της συνεδριάσεως, τη συνάντηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Κοινοβουλίου που αντικατοπτρίζει την ανάγκη συντονισμού θεσμικού όσον αφορά τα θέματα ανάπτυξης και μετανάστευσης. Η ανακοίνωση που συζητούμε είναι ένα κοινό προϊόν των δύο Γενικών Διευθύνσεων ΔΕΦΚΟ και Χομ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στις συζητήσει του Κοινοβουλίου. Όπω υπεγράμμισε συνάδελφο στην Digi Home, η παραδοσιακή προσέγγιση όσον αφορά τα θέματα τη μετανάστευση και τη ανάπτυξη που ακολουθήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι ανεπαρκές για να αντιμετωπιστούν πραγματικά και εξαντλητικά τα θέματα του αντικτύπου της μετανάστευσης επί των αναπτυσσομένων χωρών. Η ανακοίνωση ακολουθεί την κατεύθυνση που πάει πιο μακριά από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα αν θέλουμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό και να λάβουμε υπόψη όλο το δυναμικό της μετανάστευσης σαν παράγοντας διευκόνησης ανάπτυξης. Χρειάζεται καλύτερη στόχευση όσον αφορά τι συνέπειε επί της αναπτύξεως, της μεταναστεύσεως από νότο προς νότο, στο βαθμό που η ανάλυση αφορούσε βασικά την μετανάστευση που την Ευρώπη. Τώρα θα το πεδίο. Να έχουμε υπόψη αυτό που ανέφερε η συμπρόεδρο, ότι περίπου το ίμιση των διεθνών μεταναστών διαμένει σε χώρες μέσω και χαμηλού εισοδήματος και 80% των Αφρικανών μεταναστών ε, ζουν σε μια άλλη Αφρικανική χώρα. Η μετανάστευση έχει θετικές και συνέπειες όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των ανεπτυσσομένων χωρών που είναι και χώρες προορισμού. Όμως πολλές από αυτές τις χώρες δεν έχουν συνεκτικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη μετανάστευση προς δικό τους όφελος και την προστασία, την επαρκή των μεταναστών εργαζομένων, των μεταναστών εν γέννη και των μεταναστών εργαζομένων πιο ειδικά. Η μετανάστευση νότος-νότος έχει σημαντικές συνέπειες για τις χώρες προέλευσης, Προς χάρη 20 με 30% όλων των χρηματοπιστωτικών μεταφορών γίνονται μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών, Μέχρι τώρα αυτό δεν το είχαμε αναλύσει επαρκώς. Ε, η συζήτηση όσον αφορά τη μετανάστευση και ανάπτυξη επίσης ίσως τόνιζε περιβολικά την οικονομική συνέπεια της μετανάστευσης χωρίς να αναλύει επαρκώς τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Κάποια θέματα πιο συγκεκριμένα και πιο ειδικά διερευνήθηκαν επαρκώς όπως η σχέση μεταξύ αλλαγής του κλίματος και μετανάστευσης, ε, αστικοποίηση, αστιφιλία και μετανάστευση και σχέση μεταξύ ανάπτυξης και προσφύγων. Ε, λόγω αυτού ε, κάνουμε στην ανακοίνωση προτάσεις για να εξασφαλίσουμε πιο φιλόδοξη και ευρία προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Να μην εξετάζονται αυτά μόνο σε διαλόγους υψηλού επίπεδου, αλλά να εφαρμόζονται αυτές οι προσεγγίσεις και στις πολιτικές συνεργασίες. Οι προτάσεις που γίνονται ισχύουν και για την ατζέντα, για την αλλαγή και, και το όλο φάσμα της ανάπτυξης και μετανάστευση. Τα δύο πολιτικά πλαίσια αναφοράς που έχουμε. Η ανακοίνωση θα εξασφαλίσει ότι το πολιτικά πλαίσια είναι συμπληρωματικά ότι δίνουν ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεργασίας ευρωπαϊκής όσον αφορά προτεραιότητες για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Υπάρχουν επίσης και προτεραιότητες συμπληρωματικέ στα πλαίσια και στο πρόγραμμα για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Έτσι βελτιστοποιείται μεγιστοποιείται ε, η συνέπεια της ανάπτυξης όσον αφορά την ανάσταση προς την Ευρώπη. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς, όπως τη μείωση του κόστου των, της μεταφοράς των ε, εμβασμάτων. Ε, γίνονται προτάσεις ούτω ώστε η μετανάστευση να αντιμετωπίσει στα πλαίσια της συνεργασίας της αναπτυξιακής με εξαντλητική προσέγγιση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να εξετάσουμε όλες τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πτυχές που μπορούν να λάβουν οι διάφορες μορφές της μεταναστεύσης και διάφορες μορφές που μπορεί να λάβει ούτως ώστε να έχει συνέπειες όσον αφορά την ανάπτυξη οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο στις χώρες που είναι χώρες προέλευσης και προορισμού ε, οι οποίες είναι χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Χρειάζεται καλύτερη στόχευση όσον αφορά τη συμπερίληψη της μεταναστευτικής διαστάσεως, κάτι που κάνουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει ανάγκη να συμπεριλάβουμε τη μετανάστευση σαν, τη θεωρήσουμε σαν πρόκληση και σαν δυνατότητα και ευκαιρία για την ανάπτυξη και να τη συμπεριλάβουμε στις πρωτοβουλίες μας για συνεργασία όσον αφορά τα γεωγραφικά μέσα. Όποτε αυτό είναι εφικτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητούμε η μετανάστευση να είναι ένα θέμα εστιακό, αν δεν γίνεται σε επίπεδο ε, χωρών, αυτό όμως μπορεί να γίνει σε επίπεδο περιφερειών. Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε οι χώρες εταίροι να συμπεριλάβουν αυτή τη μεταστευτική διάσταση και η πρώτη φάση είναι να φροντίσουμε ούτω ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν την πραγματική αξία της μετανάστευσης και την εντάξει στις πολιτικές τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να βοηθούμε τις χώρες εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θα φροντίσουμε το ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την ενίσχυση της μεταστατικής διαχείρισης και δικυβέρνησης κάτι που κάνει και όσον αφορά τα θεματικά και γεωγραφικά μέσα. Και αυτό για να καλύψουμε όλους τους τομείς μετανάστευσης. Μετανάστευση για λόγους ε, εργασίας και διαχείριση των συνόρων. Όλο το φάσμα. Ένα λεπτό. Είσαστε καλός, πολύ καλός. Βλέπω να κινείτε το σφυρί σας και ανησυχώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε ότι η εφαρμογή όλων αυτών των υποχρεώσεων που είναι φιλόδοξε, απαιτεί πολιτικού προσανατολισμού επί διαφόρων αμεληθέντων μέχρι τώρα θεμάτων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκολύνουμε τι σχηματοστατικές μεταφορέ, να βοηθήσουμε τι χώρε μέσω και χαμηλού εισοδήματο προορισμού, να ενισχύσουμε τη κυβέρνηση και τη διαχείρισή του με το ροών και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών με τι ευρωπαϊκέ χώρε, να βελτιωθεί η κατανόηση του φαινομένου θα πρέπει οι πρόσφυγες να ενταχθούν στα αναπτυξιακά προγράμματα και όλος ιδιαιτέρως εκείνους που ε, έχουν παγιδευτεί. Θέλουμε να βγούμε από την ανθρωπιστική προσέγγιση και να δούμε πώς οι πρόσφυγες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ε, των διαφόρων κοινοτήτων υποδοχής Πρέπει να βαθύνουμε τι γνώσει μα όσον αφορά τι οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε τη μετανάστευση και να βρούμε τη σχέση μεταξύ αλλαγή του κλίματο, επιδείνωση περιβαλλοντική, ε, σύμφωνα με αυτά που αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του έγγραφου εργασία μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Θεμάτων. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σταματώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Είναι προφανές ότι έχουμε υπερβεί το χρόνο της διερμηνίας. Τους ευχαριστούμε για τη γενοδορία τους, για το συμπεριλημματικό χρόνο που μας έδωσαν. Σας παρακαλώ να ολοκληρώνετε, διότι καταναλώσαμε ένα λεπτό, ήδη και έχουμε να ακούσουμε και τον κύριο Χέμιγκουε. Τελειώσατε? Α, ευχαριστώ. Ο κύριος Χέμιγκουε, λοιπόν έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για την χρονική πίεση. Ευχαριστώ τους διερμηνείς που μας δίνουν και κάποια λεπτά παραπάνω για να συνεχίσουμε. Ορίστε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να αναφέρω ακροθυγώς κάποια σημεία και προσπαθήσω να παραμείνω στο χρονικό διάστημα στη διαθέσή μου. Σαν διεθνή οργανισμό με παγκόσμια εντολή και με που επηρεάζει η μετανάστευση, έχει γνωστή μετανάστευση, προετοιμάζουμε τον διάλογο υψηλού επίπεδου και κατόπιν αιτήματο τη Γενική Συνελεύσεω του ΟΗΕ και των 150 100 μελών το φορέ εκτελεστικό στο ΙΕ εξέδωσε μια απόφαση τον Απρίλιο του 2012 που ζητά από τα ΙΕΜ και του διάφορου άλλου φορείς να προετοιμάσουν σε συνεργασία με την παγκόσμια, ομάδα την παγκόσμια για τη μετανάστευση διάφορε συστάσει όσον αφορά τη μετανάστευση και την προετοιμασία για την Σύνοδο Κορυφή για το υψηλό επίπεδο διάλογο του 2013 και δράτω με τι ευκαιρίε για να αναφέρω κάποιε από τι σκέψει μα όσον αφορά τα σενάρια που μπορεί να ακολουθήσει ο διάλογος ψηλού επίπεδου. Καλωσορίζω την πρόταση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή τη όσον αφορά τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του αναπτυξιακού τη μετανάστευση σε ένα έγγραφο που ευθυγραμμίζεται με τις έννοιες που έχουμε στο έγγραφο τοποθέτηση για τη συζήτηση ψηλού επίπεδου του IOM που ολοκληρώθηκε αυτό το έγγραφο το Φεβρουάριο φέτος. Η μετανάστευση έχει δυναμικό στον την ανάπτυξη και θετικά αποτελέσματα, όμως δεν μπορούμε να τα εγγυηθούμε. Η μετανάστευση ε, ε, ε, συμπεριλαμβάνεται στην ανάπτυξη, αλλά δεν είναι κάτι αποκλειστικό που οδηγεί στην ανάπτυξη και οι μετανάστες μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη, αλλά δεν είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη. Όσον αφορά τον τόπο μετανάστευση, όσον αφορά την παγκόσμια εξέλιξη, η πρόκληση είναι να βελτιώσουμε την, τον χειρισμό σε τοπικό και εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το χειρισμό των μετασταθμικών ροών και να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές, τις δημογραφικές, τον ανταγωνισμό για τις ε, γνώσεις και δεξιότητες, την ποικιλομορφία, ανισότητες, κοινωνική συνοχή, αλλαγή του κλίματος, ανθρωπιστική κρίση, να τα βάλουμε όλα μέσα. Λοιπόν, το IOM συνεργάζεται στενά με την ομάδα την Παγκόσμια Μετανάστευση και θεωρούμε ύψη τη σημασία και εμείς και οι εταίροι μας του ΟΗΕ να βελτιώσουμε το συντονισμό μας και να το κάνουμε αυτό με έναν καλύτερο τρόπο, ώστε να πάρουμε και εντολή τελικά από την ομάδα υψηλού επίπεδου. Επίσης υποστηρίζουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη όπου όπως γνωρίζετε ε, τελεί υπό Σουηδική Προεδρία και είναι κάτι που υποστηρίζουμε. Εν κατακλείδη. Ο διάλογος του Λίου του 2013 είναι σημαντική δυνατότητα για να βελτιώσουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης. Λοιπόν, θέλουμε να λάβουμε υπόψη την προστασία των μεταναστών Λοιπόν, προτείνουμε λοιπόν τα εξή για τη συζήτηση ψηλού επίπεδου. Βασικά σημεία για μια πλήρη ατζέντα για να ευνοήσουμε και τις χώρες και τους μετανάστες. Και να δούμε τι γίνεται και με την ανάπτυξη σχέση με τη μετανάστευση. Να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες και να βελτιώσουμε τις θετικές. Προτείνουμε έξι σημεία. Βελτιωμένη δημόσια αντίληψη της μετανάστευσης, κάτι που δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως νομίζω ότι είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Πρέπει να εξεταστεί η αντίληψη, να υπάρξει θετική αντίληψη μετανάστευση, από τον κόσμο. Δεύτερο, στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών να μπει η μετανάστευση, καλύτερο σχεδιασμό ευθύ εξ αρχή, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα για του παράνομου μετανάστε, διαχείριση τη μετανάστευση σε περιπτώσει κρίση, μια εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την κρίση στη όπου βλέπουμε επίση και το Μαλί να εντάσσεται εκεί και είναι και αποτέλεσμα σε κάποιο βαθμό των στην Λιβύη. Θα πρέπει να διαμορφώνουμε πολιτική βάση των γνώσεων για την μετανάστευση, να συλλέγουμε στοιχεία και τέλος εξισωματικό να προωθήσουμε συνοχή των πολιτικών και θεσμική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χέμι μου, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, σίγουρα ε, πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα πρέπει να μιλάμε πιο συχνά για την μετανάστευση σε σχέση με την ε, ανάπτυξη. Επομένως ε, να γίνει πολλή έρευνα ακόμα ε, στην μετανάστευση μεταξύ χωρών του Νότου. Θα πρέπει αυτή να γίνεται προς όφελος όχι μόνο των χωρών που εμπλέκονται αλλά και προς όφελος των ατόμων. Και ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις κατευθύνσεις του UNHCR και του IOM. Ευχαριστούμε την κυρία Κέλλερ. Σύντομη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Αν όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρόζενμπεργκ, την κυρία Μπουκάτ και τον κύριο Χεμιγουέι. Και ασφαλώς την κυρία Κρέτου που εκπροσωπεί την ε, ε, Επιτροπή ΔΕΒΕ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.